Ja, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, συγγνώμη για την καθυστερημένη έναρξη της συνεδρίασης. Υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας. της ε, Προέδρου δεν θα μπορέσει να έρθει, αλλά ούτε κι εγώ κατάφερα να έρθω νωρίτερα, γιατί είχα ένα ραντεβού το οποίο δυστυχώς δεν μπορούσα να ακυρώσω. Σας παρακαλώ συγχωρήστε λοιπόν την καθυστέρηση για αυτό το μισάωρο. Δι... Διότι παρά όλες, παρά τις προσπάθειες της γραμματείας δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα. Πάμε λοιπόν στο σημείο 31 που αφορά στο, στην έκθεση του κυρίου Ντερόσα που αφορά στο μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Θα έχουμε λοιπόν την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Έχετε το λόγο κύριε Ντερόσα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Προφανώς ε, δεν είναι δικό σας ε, λάθος ε, που καθυστερήσαμε τόσο πολύ, συμβαίνουν αυτά ενίοτε. Αυτή η έκθεση έχει ως αντικείμενο το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Υπάρχει ευρεία συνένεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι στην καρδιά του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Επίσης, αναγνωρίζετε ότι ακόμη δεν τα έχουμε καταφέρει τέλεια, δηλαδή πώς συνεργάζεται η Ένωση με τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες ως καθολικές υπηρεσίες, χωρίς να σχετίζονται με το εισόδημα κάποιου, παραδείγματο χάρη. Είναι απαραίτητε για τους χρήστες αυτές οι υπηρεσίες και απαραίτητε και για τις ε, ε, μικρές ε, επιχειρήσεις, για την ποιότητα ζωής των πολιτών. Αυτό ε, έχει στοιχειοθετηθεί από διάφορες μελέτες ε, του Ιδρύματος Eurofound, ε, δηλαδή του Ιδρύματος για τις Συνθήκες Διαβίωσης και Εργασίας. Είναι σημαντικό όταν εξετάζουμε αυτό το θέμα να λαμβάνουμε υπόψη το επίπεδο στο οποίο έχουν φτάσει οι εξελίξεις ε, και ναι, να αναζητήσουμε έναν τρόπο ώστε να παρέχονται με πιο αποτελεσματικό τρόπο αυτές οι υπηρεσίες. Όσο καιρό είμαι εγώ στο Κοινοβούλιο και σίγουρα πολύ πριν από μένα, ε, ε, συνεχίζεται αυτή η συζήτηση των ε, υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Αυτές οι υπηρεσίες καλύπτουν οικονομικές υπηρεσίες και μη οικονομικές υπηρεσίες. Είναι δύο υποδιαιρές που υπάρχουν. Οι κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος ανήκουν και στις δύο κατηγορίες, και στις οικονομικές και στις μη οικονομικές υπηρεσίες. Και σίγουρα θα υπάρξουν διαφορές και αντιδικίες ε, όταν κληθούμε να χαράξουμε τη διαχωριστική γραμμή. Μάλλον ε, κατά περίπτωση θα πρέπει να κρίνουμε. Τον Ιούνιο του 2007 με την έκθεση Φερέιρα είναι η τελευταία φορά που συζητήσαμε αυτό το θέμα ε, και σε εκείνη την έκθεση η πιο βασική πρωτοβουλία κατ' ήταν η πρόταση για σύσταση ενός φόρουμ ώστε τακτικά να ε, αναθεωρούμε την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ε, πριν από λίγους μήνες υπό την αιγίδα της Βελικής Προεδρίας συναντήκαμε με το φόρουμ αυτό και προέκυψαν εξάλλου και 15 συγκεκριμένες συστάσεις από το φόρουμ σχετικά με την πρόοδο που πρέπει να σημειωθεί για τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Προσπάθησα να ενσωματώσω αυτές τις συστάσεις και στη δική μου έκθεση. Επίσης έλαβα υπόψη τις απόψεις ε, των εμπλεκομένων φορέων, ε, μιας ευρείας δέσμης ε, φορέων, κοινωνικοί εταίροι, αλληλασφαλιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις, προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη την άποψη όλων των ενεχόμενων φορέων. Μας βοηθάει αυτό πολύ στην εκπόνηση των προτάσεών μας. Ε, το σημαντικό είναι να είμαστε ρεαλιστές. Ε, εγώ δεν θέλω να προκύψει διχογνωμία στο Κοινοβούλιο για αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες. Εξάλλου σας είπα, υπάρχει ευρεία συνένεση. Όχι ομοφωνία, αλλά ευρεία συνένεση όλα τα θεσμικά όργανα, με όλα τα θεσμικά όργανα εξάλλου και με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το στόχο που επιδιώκουμε για τις ε, κοινωνικές υπηρεσίες. Τώρα, ε, ισχύουν με τις νέες μάλλον περιστάσεις, ε, με την κρίση στον τραπεζικό τομέα και στο χρηματοπιστωτικό τομέα που έχει πλήξει την οικονομία μας, αλλάζουν τα δεδομένα και επηρεάζονται και αυτές οι υπηρεσίες, οπότε θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο ώστε να υπερπηδήσουμε αυτό ε, το εμπόδιο και να λύσουμε αυτό το γόρτιο δεσμό αν θέλετε. Με στην έκθεση προσπαθώ να εντοπίσω τρόπους αντιμετώπισης του, της νέας κατάστασης. Άλλη σημαντική αλλαγή, η διατάξη της συνθήκης Λισαβόνας. Εκεί τονίζεται ότι ε, κατευθυνόμαστε προς μια κοινωνική οικονομία, προς περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, προς εκπόνηση όλων των πολιτικών λαμβάνοντας υπόψη την ε, κοινωνική διάσταση. Στο άρθρο 3 προφανώς περιγράφεται η Ευρώπη ε, που επιθυμούμε να οικοδομήσουμε μια αποτελεσματική ε, οικονομία με κοινωνική διάσταση. Ε, ε, χρειαζόμαστε και τα δύο. Το άρθρο 14 προβλέπει την δυνατότητα να ψηφιστεί ένας κανονισμός πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος και κατόπιν έχουμε το πρωτόκολλο 26 όπου προβλέπεται ότι οι υπηρεσίες αυτές επαφίονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ε, κρατών μελών εκείνα πρέπει να ορίσουν ναι, ε, τι εστί ε, κοινωνική υπηρεσία, οικονομικής δραστηριότητας, μη οικονομικής δραστηριότητας και ούτω καθεξής. Άλλα στοιχεία τώρα της συνθήκης επηρεάζουν αυτά τα δικαιώματα. Παραδείγματος χάρη για τις κρατικές προμήθειες ε, τακτικά γίνονται προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μια αντιδική ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις, ε, και μια αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή ε, ανάμεσα σε έναν νοτά και μια εταιρεία για τον τρόπο παροχής κάποιων κοινωνικών υπηρεσιών. Κατά τη γνώμη μου προέκυψαν από αυτές τις προσφυγές καλές και κακές αποφάσεις. Η απόφαση Χάλπμαρκ, όπου βάσει της οποίας ε, ετέθη το όριο, το κατόφλι για την κοινωνική στέγη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καλής απόφασης. Ε, περιγράφουμε την κοινωνική υπηρεσία, αν πρέπει να είναι καθολική υπηρεσία αυτή της κοινωνικής στέγης, αν θα παρέχεται μόνο στους απόρους κτλ. κτλ. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που πρέπει να ρυθμίσουμε σε σχέση με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Ε, προσπάθησα μέσα στην έκθεσή μου, όπως σας είπα, να είμαι ρεαλιστής. Φερρυπίν, δεν ενσωμάτωσα, ενώ είχα τη φυσική τάση να το κάνω ομολογουμένος και θα το δείτε στην εταιρεολογική μου έκθεση, δεν συμπεριέλαβα μία ε, πρόταση για μία οδηγία πλαίσιο για τις κοινωνικές ε, υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Μπορούμε να κάνουμε μία μεγάλη συζήτηση, αν θέλετε, για αυτό το θέμα. Θα είναι και συναισθηματικά φορτισμένη και μπορεί να κλείνει η πλάση προ οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αλλά ε, δεν είναι αυτό το σημαντικό για μένα. Θέλουμε ποιοτικέ, αποτελεσματικέ ε, κοινωνικέ υπηρεσίε γενικού ενδιαφέροντο. Ναι, μένα, αλλά εγώ προσπάθησα να εστιάσω την προσοχή μου στα ζητήματα που πρέπει να προσδιοριστούν και να ρυθμιστούν για να καλυφθούν οι ανάγκε των κοινωνικών εταίρων. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω απαντήσει στα ζητήματα που αφορούν άμεσα ε, του κοινωνικού εταίρου. Ε, δεν ισχυρίζομαι ότι είναι τέλεια η έκθεσή μου και προφανέστατα θα θα και τροπολογίες ε, από τους συναδέλφους ε, στο μέτρο που εγγράφονται στα πλαίσια της συνθήκης, γιατί η συνθήκη είναι το έρισμα ε, όλων των πρωτοβουλίων και δραστηριοτήτων μας. Κάτι άλλο στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω τώρα. Έγινε το τρίτο φόρουμ για τις κοινωνικές ε, υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος ε, και μία από τις προτάσεις μου είναι ε, να συγκαλέσουμε σε δύο χρόνια τέταρτο φόρουμ που θα διοργανώνει η Επιτροπή μας, γιατί είμαστε βασικοί παράγοντες στην όλη διαδικασία ε, φυσικά δεν είναι η τέλεια λύση, ούτε είναι θέσφατα αυτά που λέω. Θα ε, βρούμε μια λύση. Το σημαντικό είναι να ε, τονώσουμε την δυναμική που υπάρχει για να σημειωθεί πρόοδος σε όλους αυτούς τους τομείς. Εξάλλου οι συνάδελφοι βουλευτές θα εντοπίσουν πού πρέπει να σημειωθεί η πρόοδος. Επίσης, σε μια task force, μια ομάδα εργασίας όπου θα εκπροσωπούνται όσο το περισσότερο περισσότεροι φορεί γίνεται, ε, ε, δηλαδή οι οργανώσει κοινωνία των πολιτών, οι Γενικέ Διευθύνσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, οι αρχέ τοπική αυτοδιοίκηση, οι περιφερειακέ αρχές, ε, υπάρχουν πάρα πολλέ ε, αντιπροσωπευτικέ ε, οργανώσεις και νομίζω ότι όλοι πρέπει να εμπλακούν σε αυτό το διάλογο. Εν πάση περιπτώσει η αρχή είναι να έχουμε ένα διαφανή μηχανισμό ο οποίος θα βασίζεται στην αρχή της διαφάνειας ε, για να κατοχυρώσουμε την ισότιμη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, να ε, οριοθετήσουμε τα ζητήματα προ επίλυση και να υπάρχει αλληλεπίδραση ούτω ώστε να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος. Αυτή η ομάδα εργασία κατόπιν ε, θα υποβάλει έκθεση στο τέταρτο φόρουμ σε δύο χρόνια για την πρόοδο που θα έχει σημειωθεί ε, δεν είναι ιδεολογικό το θέμα για μένα, ε, η στο εμπαρόδο. Προσπαθώ να βρω τρόπους ώστε ε, να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών που χρειάζονται αυτές οι υπηρεσίες, να καλυφθούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες. Δεν υπάρχει επιχείρηση που δεν εξαρτάται από μια υψηλής ποιότητας εκπαιδευτική, παραδείγματο χάρη, υπηρεσία. όλοι χρειάζονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον τομέα τη υγεία, στον τομέα των δημοσίων μεταφόρων, σε ένα σωρό τομεί ε, που έχουν καθοριστική σημασία. Σήμερα το πρωί σε μια συνεδρίαση είπε κάποιο ε, ότι οι ιδιωτικέ επενδύσει είναι ε, ο κινητήρα τη ανάπτυξη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό σημαντικό είναι, δεν αντιλέγω, αλλά οι κοινωνικέ υπηρεσίε ε, είναι το καύσιμο, αν θέλετε, τότε που, με το οποίο λειτουργεί αυτό το όχημα, του οποίου ο κινητήρα είναι η ανάπτυξη. Ε, και νομίζω ότι δεν θα το αμφισβητήσει αυτό κανείς. Δεν υπάρχει διαμάχη, ε, ε, δεν είναι αντικρώμενες έννοιες οι ιδιωτικέ επενδύσεις, δηλαδή και η ιδιωτική δράση από τη μία και οι καθολικές υπηρεσίες από την άλλη. Οι επιχειρήσει δημιουργούν θέσει απασχόληση, μα δίνουν τα προϊόντα, τα χρειάζεται αυτά η κοινωνία, αλλά χρειάζεται και τι κοινωνικέ υπηρεσίε. Κατόπιν, μια τελευταία αναφορά στο εθελοντικό πλαίσιο ποιότητας που έχει ήδη αρχίσει να ε, διαμορφώνεται. Θα δούμε πώς μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω. Ε, σε θελούσια βάση πάντως θα πρέπει να λειτουργεί. Υπάρχουν ε, διαφορετικές ποιε απόψεις σε σχέση με την ε, ποιότητα των υπηρεσιών, το επίπεδο ποιότητα στο οποίο πρέπει να αποσκοπούμε και μην ξεχνάτε ότι σε κάποιε χώρε υπάρχουν υπηρεσίες σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με άλλες, άρα θα έχουν ε, και άλλους στόχους. Επίσης να λάβουμε υπόψη τα κοινωνικά κριτήρια κατά την παροχή των ε, κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος, όχι μόνο να μα απασχολεί η ποιότητα μάλλον να μας απασχολεί ποιότητα και για αυτούς που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και για τους παρόχους των υπηρεσιών. Επίσης υπάρχουν υπηρεσίες που παρέχονται από το δημόσιο και άλλες από τον ιδιωτικό τομέα. Όταν υπάρχει εξωτερική ανάθεση μιας υπηρεσίας σε έναν ιδιωτικό πάροχο, πιστεύω ότι πρέπει να προβλέπεται απέτηση να πληρούνται και κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια. Ε, εν γέννη, ε, αυτό είναι το περιεχόμενο, αυτός είναι ο στόχος εκθεσής μου. Ελπίζω να γίνει ζωντανή συζήτηση και προσβλέπω σε μια ευρία συνένεση ε, για το θέμα αυτό. Το χρειαζόμαστε για να προοδεύσουμε και να επιδείχουμε ποιοτικέ υπηρεσίε, ε, κοινωνικέ υπηρεσίε γενικού ενδιαφέροντος που θα εξυπηρετούν στο μέλλον του πολίτε τη Ένωση. Σα ευχαριστώ πολύ. Εμεί σα ευχαριστούμε. Κύριε Σιγητά. Και περνάμε τώρα στις συμβολές των σκιωδών εισηγητών. Κύριε Ρεγκίνα Παστός, είναι η πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και σαφέστατη για τις ε, θέσεις που περιέγραψε μόλις ο εισηγητής μας. Συγχαρητήρια εξάλλου. Κύριε Ντερόσα, για την εργασία σας και την, ε, το σχέδιο έκθεσης που μας παρουσιάζετε. Αυτή η ρεαλιστική προσέγγιση στην οποία επιμείνατε ε, καθ θυσιχάζει τις ε, ανησυχίες ε, που υπάρχουν και κατευνάζει την ε, οποιαδήποτε ιδεολογική συζήτηση γίνεται για τα ζητήματα των κοινωνικών υπηρεσιών και έτσι πιο, με πιο ομαλό, με πιο εύρυθμο τρόπο μπορούμε να συνεχίσουμε το διάλογο κυρίως σε μια εποχή όπου έχουμε πληγεί από την οικονομική κρίση και φυσικά πλήττονται και οι ίδιες οι κοινωνικές υπηρεσίες από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Είναι έχουν βασική ε, θεμελιώδη σημασία αυτές οι υπηρεσίες για την εδαφική και κοινωνική συνοχή. Γνωρίζουμε ότι αυτές οι υπηρεσίες είναι κομμάτι της καθημερινότητας ε, των ε, πολιτών στον τομέα της υγείας, των μεταφορών, της υδροδότησης, σε πάρα πολλούς τομείς. Επηρεάζεται άμεσα η αξιοπρέπεια των πολιτών, το επίπεδο διαβίωσής τους, η προστασία που τους παρέχουμε, όλα αυτά είναι συνάδελφοι Τη ποιότητα ε, των ε, κοινωνικών υπηρεσιών και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι σε αυτό το τομέα ε, τα κράτη-μέλη και οι περιφερειακές αρχές και όλες οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης εμπλέκονται άμεσα σε επίπεδο κρατών μελών. Ε, οι υπηρεσίες αυτές επαφείται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. άρα Ε, μάλλον λόγω του ότι θα πρέπει να είναι όσο δυνατόν πλησιέστερο στον πολίτη γίνεται αυτές οι υπηρεσίες. Άρα δεν επιθυμούμε να έχουμε ευρωπαϊκή σε εισαγωγικά παρέμβαση. Χρειαζόμαστε όμως μια σαφή νομική βάση ούτω, ώστε να είναι διαφανής η όλη διαδικασία. Αλλά κατά τη γνώμη μας δεν χρειάζεται οδηγία πλαίσιο. Ε, σε επίπεδο ένωσης, διότι αυτό μπορεί να ανατρέψει ε, τους κανόνες ε, οργάνωσης και χρηματοδότησης αυτών των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Α, θέλουμε να μεριμνήσουμε ώστε να είναι ποιοτικέ και προσβάσιμες αυτές οι υπηρεσίες. Αντιλαμβανόμαστε ότι ε, ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε επίπεδο κράτους μέλους και σε επίπεδο περιφερειακών και τοπικών αρχών και όχι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίοδο κρίσης ε, και εξάλλου ο εισηγητής μας ο κύριος Ντερόσα το τόνισε αυτό, ε, ζούμε, ισχύουν ε, νέα δεδομένα σε σχέση με την κατάσταση του 2005 όταν ε, εκπονήθηκε η έκθεση Φερέιρα. Έχουμε την κρίση και άρα πρέπει να προσέξουμε για να παράσχουμε με ικανοποιητικό τρόπο αυτές τις υπηρεσίες, αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα, η κοινωνική οικονομία της αγοράς, στη, την οποία επιδιώκουμε για να εξέλθουμε και από την κρίση και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 14 της ε, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωση καθώς και το πρωτόκολλο 10 ε, ως νομικά ερίσματα για τι νέε διατάξει. Δεν πρέπει να έχουμε προκαταλήψει σε καμία περίπτωση σε σχέση με τον εθνικό τρόπο οργάνωσης αυτών των υπηρεσιών ε, είτε παρέχονται από το δημόσιο υπηρεσίες είτε υπάρχει εξωτερική ανάθεση στον ιδιωτικό τομέα να σεβαστούμε τις εθνικές παραδόσεις και να παρακολουθούμε ε, από κοντά την πρόοδο που ε, σημειώνεται ε, και να λαμβάνουμε υπόψη τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να είναι προσβάσιμες υπηρεσίες, να μην έχουμε κοινωνικό αποκλεισμό και να είναι κυρίως αποτελεσματικές αυτές οι υπηρεσίες. Επίσης, ε, μας ικανοποιεί αυτή η πρότασή σας για τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας, της ομάδας μελέτης, Task για το θέμα αυτό. Μπορούμε να συνεργαστούμε κάλλιστα μαζί σας, διότι είναι όντω ρεαλιστική η προσέγγιση σας σε μια περίοδο όπου οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα κληθούν να προσφύγουν ε, συχνότερα από ό,τι στο παρελθόν σε αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέρον λόγω της κρίσης. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ κύριε Βαστός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντερόσα για την εργασία του που συμπεριλαμβάνει όλα τα σημεία κλειδί τα οποία συζητήσαμε και στο φόρουμ για τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να προσέχουμε. Να προσέξουμε ώστε τα κράτη να μπορέσουν να εγγυθούν τη διατήρηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού για τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος και για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Πρέπει να έχουν ένα σταθερό προϋπολογισμό σχετικά. Στη συνέχεια, σχετικά με τον δημοσιονομικό φάκελο, εγώ νομίζω ότι μια φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μπορεί να βοηθήσει τα δημοσιονομικά. Θα πρέπει επίσης να έχουμε κριτήρια, ποιοτικά κριτήρια, είτε κοινωνικά είτε περιβαλλοντικά, τα οποία θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά κατά τις δημοπρασίες. Επίσης, Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αναγνωρίζει ότι οι υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος λειτουργούν, με, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, με μία λογική μη εμπορική. Δεν είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Η ποιότητα ζωής των πολιτών εξαρτάται από την ποιότητα των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. Τώρα, εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι το νομικό. Στη συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής αρχής, δηλαδή συνεργασία μεταξύ δημοσίου και δημοσίου. Και όταν μιλάω για ποιοτικά κοινωνικά κριτήρια, είναι και των συνθήκων εργασίας, η σημιστή, ε, και γιατί τίθεται εδώ το πρόβλημα μιας οδηγίας. Διότι όπως αναφέρατε, εδώ και πολλά χρόνια εργαζόμαστε γύρω από αυτό το θέμα. Ρωτώ, τι θα κάνουμε μετά την έκθεση, τι χειροπιαστό θα παρουσιάσουμε στον πολίτη, Εγώ εκ μέρους της ομάδας των Πρασίνων θα κοιτάξω να δώσω σαφείς απαντήσεις σε όλα αυτά μέσα από τις τροπολογίες που θα καταθέσω. Ευχαριστώ πολύ. Φάμπα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή που προετοίμασε ο κύριος Δελώσα δεν θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ασαφής. Θα πρέπει ξεκάθαρα να πούμε ότι η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών αυτών θα οδηγήσει οπωσδήποτε στην επιδίνωση. διακόπτη η πρόεδρος. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την διερμηνία. Vielleicht versuchen Sie einfach να ξαναρχίσετε τώρα, νομίζω ότι θα λειτουργήσει το σύστημα. Ναι, ωραία. σα ευχαριστώ. Θα ήθελα να επιστρέψω στην προσοχή σα στο γεγονό ότι η ιδιωτικοποίηση, γιατί περί αυτού συζητάμε, η ιδιωτικοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών οπωσδήποτε οδηγεί στην επιδείνωση των υπηρεσιών. Είναι χειρότερη ποιότητα και πιο ακριβές. Όταν κανένας παράγει κάποια αγαθά, ε, υπάρχουν κάποια ε, εργοστάσια που παράγουν τα αγαθά αυτά και υπάρχει η ζήτηση μεταξύ των πολιτών. Όμως όσον αφορά τις ε, καθολικές αυτές υπηρεσίες η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Δεν θα ήθελα λοιπόν η έκθεση αυτή να καταλήξει όπως όλες οι άλλες παρόμοιες εκθέσεις μέχρι στιγμής. Πρόεδρος, ευχαριστώ συνάδελφε Φάμπερ. Ελίζα Μαγόν Ζόντια έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Ντερόσα για τη δουλειά του. Είχαμε την ευκαιρία στην μόνιμη ομάδα εργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξετάσουμε αυτό το θέμα. Η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα πλούσια και αντικατοπτρίζεται εδώ και όλη η δουλειά η οποία ε, έγινε διότι συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο. Σε αυτά τα οποία είπε η κυρία Μπαστός και η Καρίνα Ντελή. Πρέπει να προσέξουμε πολύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορούμε να τα ζητάμε όλα από τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να τους πούμε ότι προσέξτε πρέπει να έχετε ισορροπημένους εθνικούς προϋπολογισμούς προσοχή αν δεν σεβαστείτε αυτή την ισορροπία τότε εμεί θα αναλάβουμε κυρώσεις όπως λέγαμε σήμερα το πρωί. Και τώρα εγώ ακούω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να δεσμευτούν να κρατήσουν ε, το επίπεδο των χρηματοδοτήσεων των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Αν εμείς θέλουμε η Ευρώπη να μας πάρει να παίρνεται στα σοβαρά από τον κόσμο, δεν μπορούμε να τα ζητάμε όλα στα κράτη-μέλη. Πρέπει να προσέξουμε. Ναι, μπορούμε να είμαστε σύμφωνοι για πραγματικές κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος οι οποίες συνεισφέρουν στον κοινωνικό ιστό είτε σε αστικό πλαίσιο είτε σε, στην ύπεθρο σύμφωνοι. Αλλά προσοχή, δεν πρέπει εμείς να αρχίσουμε να πιέζουμε, να πιέζουμε σε όλα τα επίπεδα γιατί αυτά θα στραφούν κατά των πολιτών μας αφενός και αφετέρου και στην ίδια την εικόνα της Ευρώπης. Να είμαστε λοιπόν ρεαλιστές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην εκπρόσωπο της Εκτελεστικής Επιτροπής. und η κυρία Κοντρέρα έχει το λόγο παρακαλώ. Thank you. I like first of all to... Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Ντερόσα για τόσο ενδιαφέρουσα και πλήρη έκθεση που μας επέβαλε και που κάνει μια πολύ πλήρη ανάλυση του τομέα των ε, υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Η Κομισιόν θα παρακολουθήσει με πολύ ενδιαφέρον την σχετική συζήτηση συμφωνούμε βέβαια ότι είναι ουσιαστική σημασία οι κοινωνικές υπηρεσίες για τους πολίτες της Ευρώπης. Πρέπει να οριστούν οι αρχές και οι στόχοι των οργανώσεων για τις κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες παίζουν ένα ε, ρόλο σημαντικό, γιατί απευθύνουν προς το σύνολο του πληθυσμού. Όπως ε, ο κύριος Αντόρ είπε πολλές φορές, δεν πρόκειται για κόστος, πρόκειται για επένδυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με χαρά βλέπω ότι οι ιδέες αυτές αντικατοπτρίζονται στην έκθεση και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα σημεία της έκθεσης. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η οργάνωση και η χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών είναι καταρχήν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Κομισιόν όμως βοηθάει τα κρατημένα να αργωνήσουν και να χρηματοδοτήσουμε ε, επαρκή ε, και χαμηλού κόστους ε, κοινωνικές υπηρεσίες. Καταρχήν εμείς ενώσαμε την ομάδα εργασίας για την κοινωνική προστασία αναφερθήκαν στο πλαίσιο για τις κοινωνικές αυτές υπηρεσίες και όπως είπε και ο κύριος Τερόσα θα εργαστούμε προς της εφαρμογής αυτής της εθελούσιας ε, πρόταση και του θελουσίου πλαίσιου. Έχουμε στα κράτη-μέλη προσπαθήσει να πείσουμε τις ε, δημόσιες αρχές ότι οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εφαρμοστούν στις υπηρεσίες αυτές. Και τι κάνουμε, δημοσίευσαμε το 2007 διάφορα έγγραφα, παραδείγματος χάρη στις αγορές, όπου αν έχουμε επίσης εγκαθιδρύσει οι υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες, να πάρουν απαντήσεις τα ερωτήματά τους, συνεργαζόμαστε με την τροπή Κοινωνικής Προστασίας και έχουμε νέες καθεδρίες γραμμές για τις τρεις ομάδες κανόνων που έχουν ήδη αναφερθεί. Σύντομα θα έχουν πρωτοβουλίες εκπαίδευσης για να μπορούν να εφαρμόζονται οι κανόνες πολύ πιο εύκολα. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη η στιγμή για να παίρνει υπόβολη αυτή η έκθεση, γιατί η Κομισιόν σκέφτεται το ενδεχόμενο της αναθεώρησης δύο σημαντικών εκθέσεων, δηλαδή των κανόνων για τους ε, κρατικές ενισχύσεις και τους κανόνες για τις δημόσιες αγορές. Έχουμε ξεκινήσει μια ευρέα διαβούλευση για τις δημόσιες αγορές. Εργαζόμαστε, ε, διαφερόμαστε συγγνώμη γι' αυτό πάρα πολύ να ακούσουμε τη συζήτηση εδώ. Γιατί φαίνεται ορισμένε από αυτές τις προτάσεις ήδη υπάρχουν στο κείμενο της έκθεσης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πού θα επιτευχθεί συνένεση. Μία παραστήριση θα ήθελα να κάνω και δεν θα εκπλήξει τον κύριο Ντερόσα. Είμαστε κάπως σκεπτικιστές όσον αφορά την ιδέα να υπάρχει μια ομάδα εργασίας με task force από διαφόρων τύπων ενδιαφερομένους. Νομίζουμε ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές για να δούμε τι υπάρχει. Εμείς δεν συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια και αντιπροσωπευτικότητα. θα μπορούμε εδώ να έχουμε ένα καλό βήμα για την εφαρμογή νέων κανόνων για τις δημόσιες υπηρεσίες. Υπάρχει μια ομάδα που δημοσίευσε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που την αναφέρετε στο σχέδιο της έκθεσής σας εσείς και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την εφαρμογή των νέων κανόνων και να πούμε ότι αυτή είναι κατάλληλη στιγμή για τη συζήτηση δεδομένων των καινοτομιών που θα υπάρχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρο, και εμεί ευχαριστούμε την Εκτελεστική Επιτροπή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Τεράσιο τώρα. Δεν έχω πολλά να προσθέσω γιατί νομίζω ότι όλοι θα θέλουν να επιστρέψουν στις πολιτικές ομάδες ε, και να συζητήσουν για τις τροπολογίες που θα καταθέσουν με τα χαράς ε, να σας ε, συναντήσω κατηδίαν ή να συναντηθούν οι πολιτικές μας ομάδες για να συζητήσουμε τις προτάσεις σας. Εν γέννη βλέπω ότι την χάνει καλής υποδοχή το σχέδιο έκθεσης. Ήθελα μόνο να πω ότι ούτως ή άλλως όσο καλή και αν είναι μια έκθεση πάντοτε θα υπάρχουν τροπολογίες. Αυτή είναι η φύση της ε, δουλειάς μας. Σίγουρα όμως θα καταλήξουμε σε μια συνενετική λύση χωρίς να πέσουμε στην παγίδα, περιέγραψε ο κύριος Φάλμπρ, δηλαδή να μην, ε, τελικά να μείνουμε με τίποτα, να μην, δημιουργεί, να μην ε, φτιάξουμε τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε να εξασφαλίσουμε μια προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες, ε, για τους χρήστες ε, των υπηρεσιών, ε, διότι αυτό προσδοκούν από εμά κυρίως με τη νέα συνήθη νομοθετική διαδικασία πρώην συναπόφαση. Θα τα καταφέρουμε στη συνεργασία μας με το Συμβούλιο. Θα ήθελα να καλωσορίσω επίσης τις απόψεις της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, προφανώς γνωρίζω ότι αντιστέκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ιδέα συγκρότησης ε, ομάδας μελέτης. Ε, δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό εμπόδιο αυτό. Η αρχή είναι κατοχυρωμένη νομίζω. Χρειάζεται ένας φορέας συντονιστικός για να σημειωθεί πρόοδος. και η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής δεν είναι ανοιχτή, δεν είναι διαφανής ε, δυστυχώς, ε, δεν μπλέκονται επαρκώς ε, μέσω αυτής στην όλη διαδικασία οι κοινωνικοί εταίροι. Νομίζω πρέπει να συζητούμε με τους κοινωνικούς εταίρους διότι χρειάζεται διαρκής αλληλεπίδραση για να δημιουργηθεί μια δυναμική Ε, δεν έχω κάτι με αυτούς που ε, εργάζονται στην Επιτροπή ε, Κοινωνικής Πολιτικής. Απλώς θέλω να εξασφαλίσω μια δυναμική πορεία για την πρόταση για να εκπληρωθούν τα, οι βασικοί στόχοι που έχω θέσει στην έκθεσή μου. Μπορούμε βεβαίως να το συζητήσουμε το θέμα, δεν είναι ότι αποκλείω κάποια ενδεχόμενα, παντός ε, θα πρέπει όποια λύση και αν επιλέξουμε να επικρατήσει διαφάνεια. Και κλεισμένον των θυρών τώρα να συνεδριάζει μια επιτροπή χωρίς καμία ε, αλληλεπίδραση με τους άμεσα ενδιαφερομένους νομίζω ε, δεν είναι καλή λύση, δεν είναι παραγωγική αυτή η μέθοδος εργασίας. Επίσης, στην προπασκευαστική φάση έκανα πολλές διαβουλεύσεις με κοινωνικούς εταίρους που κατέθεσαν ε, πολύ ενδιαφέροντα σχόλια. Κάποια μπορώ να τα συμπεριλάβω, κάποια όχι, αλλά αυτή είναι η φύση της διαδικασίας. Νομίζω έχετε και μια ημερομηνία να μας ανακοινώσετε τώρα για την υποβολή τροπολογιών. Η 23η Μαρτίου δεν μας μένει και πολλούς χρόνους δηλαδή. Οπότε ας αρχίσουμε να δουλεύουμε. Ναι, ευχαριστώ. Ακριβώ αυτό ήθελα να πω. Εγώ καταρχήν θέλω να σα ευχαριστήσω εσά και όλου όσου συμμετείχαν στη συζήτηση. Το χαδιάγαμε έχει σου την επόμενη εβδομάδα στις 23 Μαρτίου έχουμε την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και η συζήτηση των τροπολογιών 13 με 14 Απριλίου Εκεί θα εγκρίνουμε τις τροπολογίες αυτές 24-25 Μαΐου και προβλέπεται η έκθεση αυτή να περάσει στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Εδώ λοιπόν με την εξέταση αυτού του θέματος και περνάμε τώρα στο σημείο 32. Πρώτης ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγγητή είναι ο κ. Σουγκουριάνου, στον οποίο θα ήθελα να δώσω το λόγο. Thank you, Madam um, this report deals with an all Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το, η έκθεση αυτή αφορά ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ξέρετε ότι ολόκληρη δεκαετία η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούσε τα ωφέλη και τις προκλήσεις της νέας αγοράς με τις πέντε ελευθερίες κίνησης ε, κεφαλαίου ατόμων, υπηρεσιών, αγαθών και εργαζομένων. We are still debating. Um, uh, Και ακριβώς το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων μέχρι στιγμής έθεσε σε αμφιβολία τα επιτεύγματά μας. Μετά την ε, ανακοίνωση της Κομισιόν, τα προβλήματα που έχουν εργαζόμενοι όταν μετακινούνται για επαγγελματικούς λόγους είναι ακόμα πιο ξεκάθαρα. Δεν υπάρχουν τα μέτρα και προτάσεις για την βελτίωση της κατάστασης. Η έκθεσή μου αναφέρεται στα πιο έντονα προβλήματα και κάποιες λύσεις. Η κύρια μου ανησυχία είναι να εξηγήσω γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να φοβάται προβλήματα στο εθνικό επίπεδο are ε, Για να μην υπάρχουν εμπόδια. Δεν υπάρχει κανένα, κανένας λογικός, ε, λογική αντιμετώπιση για το θέμα αυτό. Και δεν είναι ιδεολογία, είναι μόνο θέμα οικονομικό. Η Κομισιόν το είπε και σε λεπτομέρειε πώ η κινητικότητα του, ε, των εργαζομένων είχε θετικού αντίκτυπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει λόγο να φοβούμαστε στο μέλλον την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από, από την Ανατολική Ευρώπη. Καταρχήν, γιατί υπάρχει συμπληρωματικό κόστος αν πάει κάποιος σε μια άλλη χώρα, παραδείγματο χάρη, είναι μια νέα γλώσσα, μια νέα κουλτούρα που πρέπει να αντιμετωθεί. Τα πράγματα δεν είναι λοιπόν εύκολα. Εκτός αυτού, εκείνοι που μετακινούνται δεν πάνε για να επιβαρύνουν την καινούργια χώρα. Συνήθως καλύπτουν κενά που υπάρχουν στην αγορά απασχόλησης. Οι δύο οδηγίε, 38 και 36, είναι πολύ σημαντικές και οι δύο. γιατί αντιμετωπίζουν ακριβώς τα υπάρχοντα εμπόδια για την εγκατάσταση των μελών της ε, οικογένειας του εργαζομένου και για την αναγνώριση των σχολικών και επαγγελματικών προσόντων. θετικό τρόπος αντιμετώπιση της σημερινής κατάστασης θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών. Ένα σημείο πάνω στο οποίο είχαμε ήδη συμφωνήσει σε συζητήσει με την Κομισιόν. Ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα να εξετάσω είναι ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων προβλέπει στενή συνεργασία μεταξύ της ε, νομοθεσίας για την απασχόληση αφενός και τις νομοθεσίες για την παιδεία, για την φορολογία κλπ. Αλλιώς δεν θα μπορεί να επιτραπεί πραγματικά αυτή η ελεύθερη κυκλοφορία. Δεν αναφερθώ σε ορισμένε από τι πηγέ που θα μπορούσαν να έχουν ε, επίδραση στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από το ε, στόχους του 2020. Γιατί αυτά θα πρέπει να συμπληρωθούν κατά κάποιον τρόπο στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Η επαγγελματική κινητικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική για τους στόχους διαλυκωτικότητας. Εκείνοι λοιπόν που δημιουργούν θέσει απασχόληση όπω η Ε και η επίσημη και η ανεπίσημη παιδεία θα πρέπει να έχουν περισσότερε δυνατότητε. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ποια είναι η παραγωγική μα σύμμαχη και ποιο είναι η αντίπαλή μα. Παράλογο διοικητικό άκθο παραδείγματο χάρη θα πρέπει να είναι και κάτι που θα αντιμετωπίσουμε κατά προτεραιότητα. Αυτά σε γενικέ γραμμέ. Θα θέλω ευχαρίστω βέβαια να ακούσω τι απόψει σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε λοιπόν στις κοιόδες ηγετρίες. Βιλίνε Πλικανβιτσιούτε. Έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκριάνο, τον εισηγητή μας. Υποστηρίζω το τις ε, βασικές ε, ε, γραμμές της έκθεσης του. Όλοι συμφωνούμε πως η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι μία από τις βασικές θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών της Ένωσης. Άρα δεν θα έπρεπε να υπάρχει η διακριτική μεταχείριση. Η πολίτες που μετακινούνται από το ένα κράτος ε, στο άλλο θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν τα δικαιώματά τους όπου και αν βρίσκονται και σε όποιο τομέα και αν δεν δραστηριοποιούνται. Ε, είτε μιλάμε για την παιδεία, είτε μιλάμε για την υγεία. Όλες οι ίδιες ευκαιρίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για όλους τους πολίτες και τις οικογένειές τους επίσης ε, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ε, υπάρχουν συχνά παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων γιατί πρέπει να μην εθελοτυφλούμε και να αντιμετωπίσουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Ε, ασκείται λοιπόν διακριτική μεταχείριση κατά υπηκόν άλλων κρατών μελών ε, σε ορισμένες περιπτώσεις για διαφόρους λόγους, διότι έχουν σε γλωσσικές γνώσεις, διότι δεν είναι εξοικειωμένοι με, τον, ε, με την ε, ένωμη τάξη του κράτους μέλους ε, στο οποίο εργάζονται. Οι εργοδότες μπορούν να ορισμένες φορές εκμεταλλεύονται τους εργαζομένους, δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες κοινωνικές εγγυήσεις. Εγώ το συνειδητοποίησα στη Λιθουανία όταν εργαζόμουν ε, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό που με ανησυχεί είναι η παράνομη απασχόληση ανθρώπων, η απασχόληση ανθρώπων στην ε, παραοικονομία. Η καταπολέμηση αυτή αυτή τη ε, παράνομη απασχόληση θα πρέπει να είναι το πρώτο στο καθήκον μα, διότι ε, η παραοικονομία ε, βλάπτει την οικονομία κάθε χώρο, δεν καταβάλλονται φόροι και δεν υπάρχουν τα, αυτά τα κοινωνικά εχέγγυα που θα έπρεπε να έχει ο κάθε πολίτης. Θα συμφωνήσω με τον εισηγητή όταν λέει ότι ήρθε η ώρα να συζητήσουμε εάν χρειαζόμαστε μεταβατικές περιόδους για να υλοποιηθούν οι διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία ε, των εργαζομένων. Τώρα έκπαινε η προθεσμία για 8 χώρες, αλλά συνεχίζεται για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ταυτόχρονα διάφορες μελέτες και αναλύσεις επιτροπής δείχνουν πώς ε, όποια κράτη-μέλη δεν εφήρμοσαν μεταβατικές ε, περιόδους δεν έχουν κάνει καταγγελίες για εργαζομένους που προέρχονται από νέα σε εισαγωγικά κράτη-μέλη νομίζω ότι θα ε, πρέπει να εξεταστεί αυτό το θέμα από τις χώρες που συνεχίζουν να εφαρμόζουν μεταβατικές περιόδους πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να φοβόμαστε ε, την αναθεώρηση των πράξεων προσχώρησης ε, στην Ένωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για έναν άλλο λόγο συχνά ακούμε ε, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μία ενωμένη οικογένεια και δημιουργείται συχνά η εντύπωση ότι εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά στο εσωτερικό της Ένωσης και κάποιοι πολίτες από τα παλιά κράτη-μέλη βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από ότι οι πολίτες των νέων κρατών. Ε, ε, έχω στείλει μια επιστολή στον Επίτροπο Ανδόρα και έλαβα την απάντηση πριν από λίγο καιρό και τι λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να επανεξετάσουν εφαρμόσουν ε, τις μεταβατικές τους ρυθμίσεις ε, ως προς την ελεύθερη κυκλοφορία των ε, μισθωτών, των εργαζομένων, διότι η κυκλοφορία μπορεί να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία, την κοινωνική συνοχή και σταθερότητα Αυτά τα σχόλια ήθελα να κάνω. Ε, αφήστε μου να σχολιάσω και ένα πιο πρακτικό ζήτημα. Μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι είναι εύκολο να μετακινείται κάποιος από ένα κράτος σε άλλο, στο ιστορικό της Ένωσης. Δίστανται οι απόψεις για αυτό. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. βλέπουμε κάποια αριθμητικά στοιχεία που δείχνουν ότι ένα μικρό ποσοστό των πολιτών κάθε χώρας ε, ε, διαμένουν ε, σε διαφορετική χώρα από τη χώρα προέλευσή τους. Σε μικρές χώρες όπως η Λιθουανία περίπου 100.000 άνθρωποι που του ενεργού εργατικού δυναμικού αποχωρούν και φεύγουν από την Λιθουανία για ένα μικρό ποσοστό. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τα αριθμητικά στοιχεία για να μπορέσουμε να μετρήσουμε και το όφελος που ε, αποκομίζουν τα κράτη-μέλη από αυτήν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Πιστεύω ότι όλα τα κράτη έχουν να κερδίσουν από αυτήν την ελεύθερη κυκλοφορία. Ευχαριστώ σας, ευχαριστούμε. Η κυρία Κορνέλσεν είναι η επόμενη ομιλήτρια από τους Πράσινους. Thank you. Um, I'd like to thank the rapporteur for, for this report and uh, I'm... Ευχαριστώ πολύ τον συνήθι για την έκθεση αυτή. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής ε, με την παράγραφο 14 που ζητάει την ε, διαγραφή, την εξάλληψη των εμποδίων μετακίνησης και πρέπει να αποφύγουν ότι τίποτα οδηγεί σε μια εκμετάλλευση των εργαζομένων. Και ήταν κάτι που οδηγούσε σε λευκή δουλεία. Φοβερό δηλαδή. Στην έκθεση αναφέρεται επίση ότι θα πρέπει να τονίσουμε τι θετικέ επιπτώσει τη κινητικότητα. Θαυμάσια αυτή η ιδέα. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να ελέγξουμε και τι αρνητικέ επιπτώσει των μεταβατικών μέτρων εν ώψη και της ένταξης της Κροατίας. Είμαι σίγουρη ότι η κυβέρνηση των κάτω χωρών θα ζητήσει μεταβατικά μέτρα για την Κροατία. παρόλο που αυτό δεν θα έχει και μεγάλο νόημα. Θα να σου πούμε ότι αυτή η ιδέα δεν είναι καθόλου καλή. άμα μπορέσουμε να εξαλείψουμε πολλά σημαντικά, πολλού ονοματικού φραγμούς στην κινητικότητα, καλά τα αναφέρει αυτό, αλλά μου λείπουν ορισμένα η αναγνώριση των γάμων ατόμων του ιδίου φύλου, που θα διευκολύνει τη δυνατότητα για τα ζευγάρια αυτά να εργαστούν στο εξωτερικό. Άτομα που έχουν αλλάξει φύλο δεν έχουν ε, ευκολία πρόσβαση σε έγγραφα που αποδεικνύουν την αλλαγή αυτή για να χρησιμοποιήσουν άλλη χώρα. Ε, όσον αφορά την αντιμετώπιση των εργαζομένων από άλλε χώρε, η Ολλανδία είναι πάρα πολύ άσκημο παράδειγμα. Ε, αυτοί που έρχονται από την Ρωμανία ή την Βουλγαρία θεωρούνται Πολωνοί. Τους λένε Πολωνούς και Πολωνούς είναι σαν βρισιά πια στην Ολλανδία αυτά τα πράγματα δεν επιτρέπεται να συνεχίσουν. Και επίσης είναι μια εποχή όπως αυτή που έχουμε περικοπές ε, γιατί υπάρχουν προβλήματα στα δημόσια οικονομικά. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την επιστροφή ορισμένων ατόμων στην πατρίδα τους που δεν έχουν πια δικαίωμα σε διάφορες παροχές του κράτους, παραδείγματος χάνει γιατί τις δικαιούνται πια μόνο εκείνοι που ζουν και πληρώνουν φόρους στην χώρα αυτή. Επίσης το θέμα της απώλειας του δικαιώματος ψήφου σε εθνικές ε, εκλογές, όταν έχει εργαστεί κάποιος στο εξωτερικό για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και μάλιστα σε ορισμένε χώρε μέλη είναι πολύ δύσκολο να ψηφίσει κανένα στι ευρωεκλογέ, ακόμα και αν εξακολουθεί να ζει στην Ευρώπη. Λοιπόν, θα για να προετοιμάσω κάποιε τροπολογίε για να είναι πιο πλήρε το έγγραφο. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Η Μύρη του Όνων έχει το λόγο. Okay, I use the same Um, Yes, uh, Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. Θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια. Είναι σωστά που αναφερόμαστε στους φραγμούς ε, της ελεύθερης κυκλοφορίας. Θα πρέπει όμως να έχουμε ένα βελτιωμένο κείμενο όσον αφορά την προστασία αυτών των μεταναστών. Είναι γνωστό σε πολλά κράτη-μέλη ότι τα άτομα αυτά είναι πολύ ευάλωτα, δεν προστατεύονται και καταλήγουν σε αβέβαιες ε, θέσεις απασχόλησης στην υποαγορά, αν θέλετε, της απασχόλησης. Θα πρέπει λοιπόν να είναι αξιοπρεπής η μετανάστευση, η ελεύθερη κυκλοφορία και θα πρέπει να το τονίσουμε το θέμα αυτό, ούτως ώστε οι όροι που ισχύουν για τους πολίτες μιας χώρας υποδοχής θα πρέπει να ισχύουν ήδη ίδιοι κανόνες και για τους μετανάστες. Στην Ολλανδία, ας πούμε, οι ίδιοι κανόνες, τα ίδια δικαιώματα θα πρέπει να ισχύουν για τους Ολλανδούς εργαζόμενους, όπως και εκείνους που έχουν έρθει από άλλες χώρες. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Γιατί δυστυχώ αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Και δεν είναι σωστό αυτό. Ούτε για τους μεταναστούντες, ούτε για τους άλλους που ζουν στη χώρα τους και υπάγονται μια πίεση, ε, υπόκεινται συγγνώμη σε μια πίεση όσον αφορά τους μισθούς και όσον αφορά τους όρους εργασίας. Το θέμα είναι πάντως πάρα πολύ σημαντικό για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Η Ελίζα Πεντεμοχών Ζώντια έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Γκουρεάνου. Εξαιρετική δουλειά. Που διέπεται και από κοινό Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την κινητικότητα την οποία όλοι, και όλοι χρειαζόμαστε μέσα στην Ευρώπη διότι όλοι θα κερδίσουμε από αυτό αλλά πρέπει όμως να είμαστε και ιδιαίτερα θετικοί και επικοδομητικοί γύρω από τους εργαζομένους που κινούνται στην Ευρώπη. Θα πρέπει εμείς να κοιτάξουμε η προστιθέμενη αξία Ή υπάρχουν πάλι προβλήματα με τη γερμανική διερμηνία. Θέλετε να ξαναρχίσω. Νομίζω ότι θα πρέπει η κινητικότητα των εργαζομένων να καταστεί θέμενη αξία διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τύχη κατάρτισης και θα έλεγα ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε ως νέα κατάρτιση αυτήν την κινητικότητα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει ασκήσει την κινητικότητα στον χώρο εργασίας έχει νέες ικανότητες, νέα ποιότητα, έχει ζυμωθεί από αυτή την κινητικότητα αποκτώντας νέα προσόντα. Και αυτά τα συμπληρωματικά προσόντα θα πρέπει να τα προσθέσουμε. Όχι μόνο ικανότητες για να ασκήσει κανείς την κινητικότητα, αλλά η ίδια η κινητικότητα θα πρέπει να αποτελέσει ένα μοχλό για την απόκτηση ε, επιπλέον προσόντων. Αυτό αποτελεί επιπλέον ε, μια προσιθέμενη αξία. Και δεν είμαστε στην υπερπροστασία αλλά στην αξιολόγηση. Δηλαδή δίνουμε νέα αξία στους εργαζομένους. Λοιπόν, εγώ παίρνω την ε, σκητάλη, κυρία Τζίμερ και μετά ο κύριος Ντερόζα. Ευχαριστώ. Καταρχήν, θα ήθελα ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση που υπέβαλε. Είναι μια πολύ καλή βάση κατά τη γνώμη μου για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με το θέμα και να μπορέσει να καθορίσει την θέση του το Κοινοβουλίο. Εγώ ανέλαβα την έκθεση για τον συνάδελφο Τζο Higgins, ο οποίος ήταν εισηγητής αλλά εξελέγει στην Ελλανδική Βουλή και γι' αυτό το ανέλαβα σήμερα. Θα σας πω λοιπόν μόνο τι προσπαθώ αυτή τη στιγμή να εξετάσω για την έκθεση αυτή. Θα ήθελα, εκτός από αυτά που ελέγχθησαν, να προσπαθήσω να εξετάσω τι δυνατότητες υπάρχουν για να υπάρχουν συγκεκριμένε απαιτήσει από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν ορισμένοι που είχαν εκμεταλλευτεί εξαιρέσεις μέχρι στιγμής τι θα γίνει με αυτούς. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχουν οι δυναμικές βάσεις στα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να εφαρμόσουν ότι ο ίδιος μισθός θα δίνεται για την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο εργασία. Και εδώ θα πρέπει να δούμε οι όροι αυτοί να επιβάλλονται. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο στα διάφορα κράτη-μέλη υπάρχουν οι απαραίτητες βάση στοιχείων για ε, στατιστική καταγραφή των ε, απεσταλμένων εργαζομένων ή να δούμε κατά πόσον πραγματικά πληρώνονται όπως πρέπει. Και θα πρέπει επίσης να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχει η υποχρέωση καταβολής ε, στα εκάστοτε εθνικά συστήματα κοινωνική προστασία, εάν η αποστολή αυτή γίνεται για πάνω από τρεις μήνες. Στα πλαίσια Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήθελα να υιοθετήσω μια πρόταση που υπέβαλε κάποια συνάδελφος να εξετάσετε περισσότερο το θέμα τι γίνεται με γάμους ή σχέσεις ατόμων του ιδίου φύλου κατά πόσο διασφαλίζονται τα βασικά δικαιώματα όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι απασχολούμενοι με το θέμα είδα ότι σε ορισμένε χώρες δεν αναφέρεται καν το θέμα της άρσης των διακρίσεων για πολίτες από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. απλώς αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν πια εξαιρέσει για τι χώρε που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Ε, και λένε ότι υπάρχουν όμως δύο χώρες για τις οποίες υπάρχουν πάντα ε, περιορισμοί. Και θα πρέπει να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε να μην υπάρχουν πια διακρίσεις. Γι' αυτό ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λίγες παρατηρήσεις έχω να κάνω. Είχαμε προηγουμένω τη συζήτηση για τις κοινοφελείς υπηρεσίες. Και νομίζω ότι εδώ Ε, δεν αποδίδεται τόσο ιδιαίτερη σημασία στους εργαζομένους που έχουν και οικογένεια. Δηλαδή περιμένουν να πάνε από τη μια χώρα στην άλλη για να εργαστούν και να αφήσουν την οικογένειά τους στη χώρα προέλευσης. Πώς θα λεφτεί η υπόψη το γεγονός ότι δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι ε, εργένιδες και δεν έχουν ευθύνε για οικογένεια. Αυτό ας πούμε ένα θέμα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Κοιτάξτε, εγώ προέρχομαι από την Ιρλανδία, που είναι μία από εκείνες τις χώρες που δεν είχαν προβλέψει μεταβατική περίοδο για τους εργαζόμενους από τα νέα τότε το 2004. Και γενικά είχαμε μια πάρα πολύ θετική εμπειρία. Εκατοντάδες χιλιάδων εργαζόμενοι ήρθαν από άλλα τμήματα της Ευρώπης για να εργαστούν στην Ιρλανδία. Υπήρχε όμως και μια μειοψηφία ατόμων που ήρθαν και που έτυχαν ανελέτης εκμετάλλευσης. Δεν έπαιρναν τον ίδιο μισθό που έπαιρναν οι άλλοι στην ίδια ε, εργασία. Πολλές ε, διατάξεις που ίσια νομικά δεν εφαρμόστηκαν. Παραδείγματος χάρη είχαν περισσότερα εργασιακά ατυχήματα από ότι οι άλλοι. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν μιλάμε για κινητικότητα. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν οι σωστοί έλεγχοι από τους επιθελητές εργασίας. Δηλαδή αν κάποιος έρθει από μια άλλη χώρα και εργαστεί στην εργασία κάπου αλλού, πρέπει να είναι ξεκαθαρό ότι προστατεύεται. ότι προστατεύεται κατευθύνει η ζωή του και η σωματική του αλλά δεν πρόκειται επίση να τύχει εκμετάλλευση ασίδωτη. Και βέβαια εμείς ανοίξαμε τότε την αγορά μας και ήταν καλόδοκτο για όλους και τότε είχαμε όμως περισσότερους επιθεωρητές σκύλων από ό,τι είχαμε για τον τόπο εργασίας. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι εκείνοι που θέλουν να μεταναστεύσουν από μία χώρα στην άλλη, που κινούνται από τη μία χώρα στην άλλη, δεν καταλήγουν να ζουν σε αναξιόπρεπες προϋποθέσεις. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Έχουμε εξαντλήσει τον κατάλογο των ομιλητών και πριν ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή θα ήθελε η Κομισιόν να μιλήσει ο κύριος Δημήτριος ή ο κύριος Φέρη ο Μάρκο φέρει από το τμήμα που είναι υπεύθυνο για το δίκτυο EURES, δηλαδή το δίκτυο που διευκολύνει ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Το 68 και το 83 οι νομοθέτες αποφάσισαν ναι, ε, να χρησιμοποιήσουν νομικό πλωστάσιο για να κατοχυρώσουν ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά ε, χρειάζεται και δημιουργία νέων θεσμικών φορέων στα κράτη-μέλη για να υλοποιηθούν αυτά. Ευχαριστούμε λοιπόν τον εισηγητή για το σχέδιο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και πληρέστατο. Θα κάνω από δύο σύντομα σχόλια, γιατί ε, από ό,τι κατάλαβα δεν έχουμε χρόνο. Πρώτον, να σας ενημερώσουμε ότι επεξεργαζόμαστε μεταρρύθμιση του Eures τώρα, ούτω ώστε, και αυτό ευθυγραμμίστε με την έκθεσή σα, ούτω ώστε λοιπόν να γίνει ε, οικονομικό εργαλείο το δίκτυο, δηλαδή να εξυπηρετούνται και οι ανάγκε και των επιχειρήσεων, διότι γίνεται με την κρίση. Υψηλή ανεργία έχουμε, αλλά χειρεύουν και πολλέ θέσει ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Ψάχνουν ε, υπαλλήλου με τα κατάλληλα προσόντα οι επιχειρήσει στα κράτη-μέλη και ε, θέλουμε να μετατρέψουμε αυτό το εργαλείο, αυτό το μέσο, να το ε, ε, καταστήσουμε ένα οικονομικό εργαλείο που θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε τους στόχους της στρατηγικής 2020. Δεύτερο σχόλιο, το δίκτυο EURES θα συμπεριλάβει την πρωτοβουλία που πρότεινε η Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο ένα πρόγραμμα ε, για να ε, βοηθήσει ε, την νεολαία από 18 έως 30 ετών για να βρουν θέση εργασίας και καλύπτοντας το κόστος για γλωσσικά μαθήματα, παραδείγματος χάρη, καλύπτοντας ε, το κόστος που συνεπάγεται η πρόσληψη ατόμου από άλλο κράτος μέλος. Επίσης, συζητούμε το ενδεχόμενο διεύρυνση της εταιρική ε, ε, σχέσης που υπάρχει μέσα στο Γιούρε. Προς το παρόν το Γιούρε συνεργάζεται με τις δημόσιες αρχές. Αλλά αυτό δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα πλέον, γιατί δεν πλήρων δεν ασχολούνται μόνο υπάρχουν μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ότα, ε, συνδικάτα που εμπλέκονται, πολλοί φορεί μέσα στην αγορά για την κάλυψη των ε, κενών θέσεων ε, εργασίας. Άρα θα πρέπει να τροποποιήσουμε τη φύση του εργαλείου τόσο ώστε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ και θα δώσω το λόγο τώρα στον ε, ειδικό μας για τα νομικά θέματα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εμείς από τον τομέα συντονισμού των κοινωνικών ασφαλίσεων δεν μπορούμε παρά να οικειοποιηθούμε της ανησυχίας που εκφράστηκε εδώ στην αίθουσα και να συγχωρούμε τον εισηγητή. Όπως διαπιστώσατε υπάρχουν ακόμη εμπόδια παρότι δηλαδή ε, η ελεύθερη, ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι ένα ατομικό εγγυμένο δικαίωμα βάσει της συνθήκης άρθρο 45 ο καθένας λοιπόν μπορεί να φεύγει από τη χώρα του και να ψάχνει δουλειά σε άλλη χώρα και να μην υπόκειται καμία διάκριση στους όρους εργασίας, στα, κοινων... στα φορολογικά, μισθολογικά, όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για την οικογένειά του. Είναι όλα αυτά πράγματα που τους ε, αναθέτει το κοινωνικό δίκαιο και βασίζεται στο άρθρο 45. Υπάρχει ένας κανονισμός ο οποίος επίσης αναφέρεται και είναι άμεσα εφαρμόσιμος συν δύο κοινοτικές οδηγίες. Αλλά από την άλλη μεριά διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πρακτικά προβλήματα και ο ρόλος μας είναι να μπορέσουμε να καταστήσουμε πραγματική την ελεύθερη κυκλοφορία γκρεμίζοντας αυτά τα εμπόδια Θέλουμε να καταστήσουμε πιο ορατά αυτά τα δικαιώματα τα οποία χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στους εργαζόμενους που μετακινούνται και στις οικογένειές τους και από την άλλη μεριά διερευνούμε και άλλες εναλλακτικές λύσεις ώστε στην πράξη αυτά τα δικαιώματα να ασκούνται καλύτερα. και ψάχνοντας και συμπληρώματα στην υπάρχουσα νομοθεσία. Καταρχήν του χρόνου κατά την Κομισιόν και αφού έχουμε προχωρήσει στην αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης θα χρειαστεί να εκπονήσουμε κανόνες για επιπλέον σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν συμβαδίζουμε και με το δικό σας στόχο για την ελεύθερη κυκλοφορία. Σας ευχαριστώ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που υποδεχόμαστε την Επιτροπή εδώ. Δεν είναι δική σας δουλειά να αξιολογήσετε την εργασία των βουλευτών. Εσείς έρχεστε εδώ και μας, μας διαφωτίζετε, μας φέρνετε τα φώτα σας. Και μετά οι βουλευτές είναι αυτοί που θα κρίνουν αν το μέτρο το, μέτρο της ε, ορθότητος ή μη ορθότητος και καλοσύνης της έκθεσης του συναδέλφου. Αυτά για την ισορροπία των θεσμικών οργάνων. Ο κύριος Ουρουάν. Ευχαριστώ πρόεδρε, ακούσαμε τόσα πολλά σχόλια, όλα πολύτιμα. Χαίρομαι διότι διαπιστώνω ότι καταρχήν υπάρχει ευρεία συμφωνία. Ακολουθούμε την ίδια κατεύθυνση. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Όλοι μίλησαν ε, για την ε, μη διακριτική μεταχείριση. Ε, προφανώς είναι απαράδεκτο και πρέπει να καταργηθεί. Αυτό που ονομάζουμε σήμερα σύγχρονη δουλεία είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα, είναι κάτι το υπαρκτό, αλλά είναι φθήνουσα η τάση ευτυχώς θα έλεγα. Επίσης, ε, έχουμε μια καλή περιγραφή της σημερινής ε, κατάστασης ε, και Νομίζω ότι ε, υπήρξαν οι υπερβολές και ε, αν θέλετε μία εσφαλμένη εκπροσώπηση των συμφερόντων των μετακινούμενων εργαζομένων. Τι εννοώ. Όταν έγιναν τα τεστ κόπωσης στα κράτη-μέλη, ε, και μία από τις ε, ε θεωρείται τότε η μετακίνηση των εργαζομένων, ε, απεδείχθη ότι τελικά δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις λόγω αυτής της ε, μετανάστευσης στο ιστορικό της Ένωσης και ας πάρουμε το παράδειγμα της Ιρλανδίας εργατικό δυναμικό από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία ανέπτυξε πολύ καλές σχέσεις με τους Ιρλανδούς εργαζομένους χωρίς περιστατικά, χωρίς προβλήματα ε, άλλοι πάλι τόνισαν τη σημασία που έχει η κοινωνική προστασία. Ε, κάτι άλλο που μου είπατε είναι ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να λύσουμε το, την οικονομική πτυχή του ζητήματος. Ε, δηλαδή, δεν θα πρέπει να αναγάγουμε σε, εξ αρχή σε, σε κοινωνικό αυτό το πρόβλημα. Λέτε, ας ρυθμίσουμε πρώτα την οικονομική διάσταση και μετά βλέπουμε. Είναι ευπρόσδεκτες οι παρατηρήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ε, προς την αναγνώριση αυτής της παράδοξης ε, κατάστασης όπου χειρεύουν, υπάρχουν και νέες θέσεις σε κράτη-μέλη σε περίοδο πλήρους οικονομικής κρίσης. Και αυτό νομίζω θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Μέσα στο σχέδιο έκθεσης ε, θα ήθελα να πω ότι εξαπλάγει με αυτά που έμαθα για την Ολλανδία. Ε, είναι γνωστοί ως Πολωνοί, τους ε, ονομάζουν Πολωνούς, τους ε, Ρουμάνους και Βούλγαρους επικούς στην Ολλανδία. Μας είπατε. Τι να σας πω, μου φαίνεται περίεργο. Είναι, καλή, ε, ε, είναι καλό αυτό το σχέδιο πιστεύω και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως βάση για τις ε, μελλοντικέ μας εργασίες και χάρη στη συνεισφορά σας θα έχουμε και μια πληρέστερη έκθεση. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Προθεσμία για τις τροπολογίες 22 Μαρτίου στις 12. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη ο συνάδελφος ε, Ρίτσαρντ Φάλμπρ για την εξέταση των 155 τροπολογιών για την εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής και πρόθεση των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και την κοινωνική ευθύνη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Θα ήθελα να αρχίσω με έναν ε, όχι παραδοσιακό τρόπο, με ένα τσεχικό παραμύθι. Ήταν ένας ε, σκύλος και μία γάτα και έφτιαχναν ένα κέικ. Η γάτα ε, προσέθεσε ποντίκια, ο σκύλος κόκαλα Ετοιμάστηκε το κέικ, ψήθηκε και ο κακός, ένας κακός σκύλος, πέρασε και έφαγε το κέικ και έπαθε φοβερό στο μαχόπονο. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής εμείς έχουμε ψήσει 7 τέτοια κακά γλυκά στην ε, Ένωση. Μέσα στην έκθεσή μου Ε, έχω προσπαθήσει να συμπεριλάβω πολλά στοιχεία και θα ήθελα ή δυνατόν να μην ε, ε, υποβάλλετε πολλές τροπολογίες. Θα ήθελα να ζητήσω τη βοήθεια των βουλευτών που δεν είναι παρόντες ε, σήμερα, αλλά ε, προετοιμαστείτε, θα είναι δυσάρεστη η συζήτηση μαζί μου λόγω της κέρυας ε, σημασίας του ζητήματος και της υποκρισίας που επικρατεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάποια κράτη-μέλη γι' αυτό το θέμα της εξωτερικής διάστασης κοινωνικής πολιτικής. Μα ζητείτε να απαιτούμε από μη κράτη-μέλη να εφαρμόζουν τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ενώ πολλά κράτη της Ένωσης ε, δεν εφαρμόζουν αυτά τα πρότυπα. Βεβαίω τώρα όλοι ασχολούνται με την κατάσταση στην Αφρική. Ε, η ύπατη εκπρόσωπος πήγε στην ε, Τρίπολη. Και δίνεται η εντύπωση ότι ε, με τη στάση που έχουν γενικότερα οι Ιθινούς, για να μην μπαίνουν σε συγκεκριμένα παραδείγματα, δεν γίνονται σεβαστά τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Ε, έχουν υποβληθεί τροπολογίες ε, ε, για να ε, διαγραφούν κάποια επικριτικά σχόλια σε σχέση με την εφαρμογή των προτύπων της εδώ εγώ υπηρέτησα στην Διεθνή Οργάνωση Εργασίας στο παρελθόν. Ε, και σας ε, επισημαίνω ότι οδηγίες όπως ε, η οδηγία για, τα, για το χρόνο εργασίας αντιβαίνουν σε πρότυπα της ΔΟΕ. Ε, γιατί με αυτή την οδηγία ο χρόνος εργασίας θα μπορούσε ε, και να υπερβαίνει τις 50 ώρες την εβδομάδα. Τέλος πάντων, ευτυχώς απέριψε το Κοινοβούλιο αυτό το σχέδιο και δεν θέλω τώρα να μπαίνω σε λεπτομέρειες. Πάντως, η τωρινή πρακτική των πολυεθνικών έχει ως εξή Αν αποφασίσουν οι μέτοχοι ότι δεν είναι αρκετά κερδοφόρος η επιχείρηση, μετεγκαθίσταται η επιχείρηση. Δείτε το παράδειγμα της Νόκια από τη Γερμανία. Μια μονάδα έφυγε και πήγε στη Ρουμανία. Η Dell πήγε από την Ιρλανδία στην Πολωνία και πολλές επιχειρήσεις μάλιστα εγκαταλείπουν ε, εντελώς ε, την Ένωση. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι μια φοβερή εφεύρεση όπως ε, η ευελιξασφάλεια, η ευελιξία με ασφάλεια. Είναι ένα πρόσχημα ε, ε, και είναι πάντοτε το ίδιο, απλώς βρίσκουμε καινούριου όρους κάθε φορά. Η... Πώς μπορούμε να μιλάμε για την εταιρική κοινωνική ευθύνη όταν η επιχείρηση καμία σχέση δεν έχει με τη χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Όσα έγγραφα, όσα ψηφίσματα, όσες εκθέσεις και αν εγκρίνουμε δεν θα αλλάξει έτσι, η κατάσταση. Σίγουρα ε, κάποιοι βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με το παρελθόν. Αν θέλετε να αμβλύνω κάπως τον τόνο που επικρατεί στην έκθεσή μου, μπορείτε να μου το ζητήσετε, αλλά να ξέρετε ότι θα είμαι δύσκολος συνομιλητής, ε, θα δυσκολευτείτε στις διαπραγματεύσεις μαζί μου, γιατί δεν σκοπεύω αυτή η έκθεσή μου να έχει την ίδια μοίρα με άλλες εκθέσεις επιτροπής, να κάθεται εδώ έξι μήνες και να μην γίνεται τίποτα. Εγώ θέλω να μας πάνουν στα σοβαρά και θέλω να ακουστεί η φωνή μας και αυτό θέλουμε να κάνω. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για να πω την αλήθεια, δεν θέλω να τρομ... Δεν θέλω να, να, να, να ε, διαφωνήσω με τον εισηγητή, γιατί είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνίες. Διότι μοιραζόμαστε τις αρχές και τις βάσεις ε, είναι μια κριτική έκθεση και χαίρομαι γι' αυτό γιατί έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα τα οποία τονίζει ο εισηγητής. Εγώ πάντως είμαι πολύ αισιόδοξη, 150 τροπολογίες είναι πολλές, εγώ πάντως είμαι σίγουρη ότι θα τα βρούμε. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στον τρόπο που λέει κανείς τα πράγματα. Ο εισηγητής θα λέει σίκα σίκα, οι άλλοι είμαστε λίγο πιο ευγενικοί γιατί αυτό το οποίο μας ενώνει ως αρχή είναι η διατήρηση του κοινωνικού μας μοντέλου. Πόσο μάλλον τώρα που βιώνουμε πλήρως την κρίση. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε το κοινωνικό μας μοντέλο και θα πρέπει να προσπαθήσουμε οι τρίτες χώρες να κοιτάξουν να μιμηθούν αυτό το μοντέλο και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε πολλές συμβιβαστικές τροπολογίες την επόμενη εβδομάδα. Η κυρία Ντανούτα και μετά η κυρία Τζίμερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. εγώ ίσως είμαι λίγο πιο αισιόδοξη από τον εισήγητη, παρά τη δήλωσή του και παρότι και εγώ έχω, είχα μια κακή εμπειρία σε σχέση με την εφαρμογή των κοινωνικών αυτών προτύπων από τότε που προσχώρησε η Λετωνία στην Ένωση το 2004 Είχα δραστηριοποιηθεί σε μια μη κυβερνητική οργάνωση και ασχολήθηκα με κοινωνικά δικαιώματα ε, και είδα συγκεκριμένε ε, περιπτώσεις ε, εργαζομένων από τη χώρα μου, ακόμη και πριν την προσχώρηση της χώρα στην Ένωση. Φυσικά υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, φυσικά υπάρχουν προβλήματα. Αλλά ε, δεν μπορούμε να καθόμαστε εδώ με σταυρωμένα τα χέρια αν θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Έχουμε υποβάλει 24 τροπολογίες ε, από πλευράς της ομάδας μου και μία από αυτές ε, σχετίζεται με αυτήν την διαγραφή ε, της αναφοράς στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Καλά, θα το συζητήσουμε κύριε Φάρμπρε, δεν είναι τίποτα ε, άσπρο ή μαύρο, όλα γκρίζα είναι. Θα συνεχίσουμε να συζητούμε. Προς το παρόν δεν έχουμε συζητήσει μαζί. Πάντως οι τροπολογίες μας είναι επικοδημητικές και έχουμε εντοπίσει ε, τα σημεία όπου μπορούμε να βελτιώσουμε την έκθεση. Παραδείγματος χάρη, ε, όταν μιλάτε για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες και έχουν την έδρα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης από πλευράς ευρωπαϊκών αρχών, ούτως ώστε να ενθαρρύνουμε να προκαλέσουμε τις θετικές εξελίξεις για τα κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα. Τέτοιου είδους τροπολογίες υποβάλαμε για την παράγραφο 10, για τη 13. για την παράγραφο 18 έχετε λάβει τις τροπολογίες μας πιστεύω ελπίζω πως ε, ο αξιότιμος εισηγητής θα δεχτεί τις τροπολογίες μας και θα τροποποιεί στο περιεχόμενο της έκθεσής του. Θεωρούμε επίσης ότι ένα από τα εργαλεία, ένα από τα μέσα είναι το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική εποπτεία και να επιβάλλουμε κυρώσεις μέσω αυτού του συστήματος σε χώρες ε, ε, όπου παραβιάζονται ε, οι εν λόγω κανόνες. Είναι η τροπολογία 22 που έχουμε καταθέσει. Προσβλέπουμε στη μελλοντική συνεργασία με τον εισηγητή, δεν φοβούμαστε και θα βάλουμε τα δυνατά μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κυρία Τσίμα. Ελπίζω ότι η πανηγυρία του κύριου Χαβέ δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι δεν θα πρέπει να προσθεθεί τίποτα στην έκθεση ή να τροποποιηθεί. Θα ήθελα να μπορέσουμε να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση μέσα της έκθεσης αυτής, γιατί διαβλέπω επίσης και τις αντιφάνσεις ε, σε σχέση με κάποιες τροπολογίες και θα ήταν καλό να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Το ένα το ανέφερε ο συνάδελφος Φάμπερ. για την πολύ διαφορετική αντίληψη της κοινωνικής πραγματικότητας στα κράτη-μέλη και ήθελα να πω ότι η εφαρμογή διπλών προτύπων σε χώρες στις οποίες είναι γνωστό ότι υπάρχουν δικτατορίες ή ότι υπάρχει το πρόβλημα της ε, κακές ε, διαχείρισης επειδή δεν έχουν ισχυρές κυβερνήσεις. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα πρότυπα, τα κοινωνικά, τα εργασιακά, τα, της προσθέσεις ε, και ελπίζω και οι άλλοι συνάδελφοι να προτίθενται να επιβάλλουν πιο αυστηρές κυρώσεις στην περίπτωση στην οποία δεν τηρούνται τα κοινωνικά περιβαλλοντικά πρότυπα. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα που τονίζουν την ανάγκη αυτή. Καταρχήν η συμπεριφορά του Ευρωπαϊκού Σώματος Εμπορίου στο Βιετνάμ, όπου δήλωσε στο Βιετναμεζικό Υπουργείο Εργασίας ότι θα ηρθεί και θα χρησιμοποιεί, θα εγκατασταθεί αλλού εάν η κυβέρνηση του Βιετνάμ επιμείνει να επιβληθούν ελάχιστη μισθή. Αυτό μου φαίνεται απαράδεκτη ανάμειξη στην εσωτερική πολιτική του Βιετνάμ και μια άλλη εμπειρία που έζησα και εγώ η γερμανική εταιρεία εν Group Χαλιβουργίας στην Βραζιλία παραβλέπει και καταπετά τα πρότυπα της προστασίας του περιβάλλοντος, ε, προβλέπει ένοπλες δυνάμεις για την προστασία του εργοστασίου από τους πολίτες κλπ αυτές οι επιχειρήσεις δεν τίνουν καθόλου να τηρήσουν μη δεσμευτικά πρότυπα. παρά μόνο εάν μπορούν πραγματικά να προσταθούν στη δικαιοσύνη και στις χώρες τους και για τα σχέδια αυτά να μην παίρνουν πραγματική ενίσχυση ή επιδότηση γιατί αυτό σημαίνει ότι κλείνουμε τα μάτια μας σφιχτά και σκεφτόμαστε «Ε, αυτό είναι πολύ μακριά, δεν μας αφορούν». Θα πρέπει να το πούμε αυτό ξεκάθαρα για να μπορούμε να δίνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και ως Επιτροπή αλλά και Κοινοβούλιο στο σύνολό του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φρονέλη. Θα μιλήσω δανεικά. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ δεν ήμουνα εισηγήτρια, αλλά ήμουνα στο Κάιρο πριν από δύο εβδομάδες και συνάντησα νεολίστικα κινήματα, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, συνδικαλιστές και όλοι έστελναν ένα μήνυμα λέγοντας ότι εμείς είμαστε ιδιαίτερα απαγοητευμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από ό,τι μας έχει προσφέρει μέχρι τώρα στην στην... στα πλαίσια της πολιτικής ή στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις προδιαγραφές εργασίας κλπ. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα βάζουν όλα αυτά σε ένα καζάνι. Και με ενοχλεί πάρα πολύ όλη αυτή η τάση. Στεναχωρέθηκα. Θα ήθελα λοιπόν να ανατρέψουμε αυτή την τάση και να αρχίσει ο κόσμος να αισθάνεται μία κάποια εμπιστοσύνη για μας. Όταν ξεκινάμε δηλαδή εμείς Όταν ξεκινάμε εμείς εξωτερικές πολιτικές λοιπόν θα πρέπει να συνοδεύονται όλα αυτά με συγκεκριμένα αυτά πράγματα. Λένε όλοι ότι το πρώτο πράγμα που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν συνάπτει συμφωνίες είναι να σκέφτεται πρώτο και καλύτερο, πρώτο και καλύτερο τον εαυτό της. Πρέπει λοιπόν να είμαστε κι εμείς πιο κριτικοί στις απόψεις που εκφράζουμε και να κοιτάμε να βοηθάμε τον κόσμο. Λοιπόν, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν που είναι... Α, ο κύριος Χάουιτ πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι υπάρχουν βέβαια και δυσάρεστες συζήτησεις. Συμφωνώ με τον εισηγητή όταν αφορά τα διεθνή πρότυπα εργασίας δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Γιατί έχουμε την ΕΛΟ που έχει κάποιες ε, συμβάσεις οι οποίες έχουν συμφωνήσει όλοι και πρέπει να εφαρμοστούν, εφαρμοστούν παντού. Είτε οι χώρε Νέα έχουν επικαιρώσει είτε όχι και εμείς θα δούμε πώς θα το επιβάλλουμε. Αυτό το σημείο κίνηση ίσω. Οι τροπολογίε που έχω προετοιμάσει όσον αφορά το θέμα της ε, ε, ευθύνης έχω να πω ότι συμφωνώ με τον ε, εισηγητή ότι δεν πρόκειται να φεύγουμε μια νέα ονομασία για να απομακρυνθούμε από τις βασικές αυτές συμβάσεις. Και αυτό ίσως σας εξηγήσει κάτι από τις μου είναι ότι είμαι αρκετά ευχαριστημένο για το ενδιαφέρον που υπάρχει για το θέμα αυτό. Είχαμε και στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπόριου μια έκθεση για τι ε, ε, πτυχές Τώρα έχουμε εδώ τι κοινωνικέ πτυχέ για την ε, εξωτερική πολιτική. Πάρα πολύ καλά όλα αυτά αυτό που δεν θα πρέπει να κάνουμε είναι να υποκαστήσουμε την υποχρέωση της Κομισιόν που θα υποβάλει μια ανακοίνωση, μας έχει υποσχεθεί τουλάχιστον. Ο Επίτροπος Ρογιάννη είπε και δημόσια ότι η ανακοίνωση αυτή θα υποβληθεί κατά διάρκεια του τρέχοντος έτους και προσβλέπουμε στην υποδοχή της γιατί θέλουμε να έχουμε πλήρη εικόνα. Και θα πρέπει να γνωρίσουμε και τον γνωρίζω αυτό στην Κομισιόν ότι κατά τη γνώμη μου μεγάλη επιτυχία μπόρεσαν να σκεγγραφίσουν κάποιες από τις άγουσες που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Ο Επίτροπος Μπαρινιέ ανέλαβε τις δημόσιες αυτές διαβουλεύσεις για την δημοσίευση μη οικονομικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα στα πλαίσια του πάζελ αυτού που εξετάζουμε. Και βλέπουμε ότι υπάρχει βέβαια ε, δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι τροπολογίε μου, δύο είναι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι κάποιες άλλες αφορούν την εργασία του Ντούν Ρόκη που είναι ο έκτακτος απεσταλμένος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για θέματα εργασιακής πολιτικής. Επίσης, κατά πόσο θα πρέπει Σέσαρ να ακολουθηθεί ε, να σας είπα, το θέμα είναι ότι δεν είναι αυτά τα ε, διεθνή εργασιακά πρότυπα. Αλλά για να πτύχουμε ίσως ε, μια καλή συνετική βάση με άλλες ε, πολιτικές ομάδες του ΣΕΣΑΡ θα μπορούσα να υποστηρίξω τη σχετική πρόταση. Αλλά θα ήθελα ταυτόχρονα να τονίσω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι οι δηλώσεις και συμβάσεις που υπάρχουν για τις εταιρείε θα πρέπει να εφαρμόζονται. Η τροπολογία μου 43 αναφέρεται στην ε, παρατήρηση Μπαρνιέ, γιατί πολλοί λένε ότι θα ήταν ίσως καλό να υπάρχει μια υποχρέωση ε, δήλωση των στοιχείων αυτών μέσα στα πλαίσια της, δημοσίευσης, της υποχρέωσης συγγνώμη, δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων. Και εντάξει, τέλος, ε, οι τροπολογίες μου 50, 81 και 151 αφορούν το γεγονός ότι θα πρέπει η ΣΣΑΡ που αυτή τη στιγμή ενημερώνεται ή γίνεται πιο επίκαιρη να ληφθεί υπόψη. Και μετά η τροπολογία 89 που αναφέρεται στο 151 ε, ε, ότι θα πρέπει εμείς δηλαδή να εργαστούμε από κοινού εδώ με άλλα μέλη του ΩΣΑ. Τέλος, η τροπολογία με 120 αφορά τα ευρύτερα διεθνή πρότυπα που ισχύουν. Θα θέλουμε να έχουμε benchmark στις ε, εμπορικές ε, συμφωνίες. Αυτό που γίνεται στην ε, Αίγυπτο, στην Ισία, βλέπουμε να υπάρχει μια αναγνώριση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν μπορούμε από τη μια μεριά να λέμε ότι υποστηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και από την άλλη μεριά να συνεχίζουμε το εμπόριο με χώρες που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτά. Και αν αυτό ισχύει για τη Βόρεια Αφρική θα πρέπει να ισχύει παντού. Και αυτό είναι το σημείο που καλύπτει η τροπολογία με 120. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στην Κομισιόν, θα ήθελα να κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις επειδή κατέθεσα καμιά δεκαριά τροπολογίες 16 τροπολογίες έχω εξαιρετικούς συνεργάτες ε, δεν είναι αυτός σκοπός η παραγωγή τροπολογιών αφορούν κυρίως σε αναφορές μέσα στη γνωμοδότηση Ε, λαμβάνει υπόψη, λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες που ο κύριος Χόουιτ ανέφερε για τη συζήτηση σχετικά με την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, όσο επίσης και τη δημιουργία ενός G20 για τα κοινωνικά θέματα. Εγώ πάντως ε, σημερίζομαι αυτήν τη διπλή του ανησυχία. Δηλαδή, την ανησυχία του για πράγματα που μπορεί να φαίνονται ως ε, ασυνάρτητα μεταξύ τους εδώ, δηλαδή ε, συνεχώς ε, εμείς προασπιζόμαστε τις αξίες ε, αξιοπρεπούς εργασίας, καλύτερες συνθήκες ζωής κλπ. Και βλέπουμε λοιπόν εμείς τι γίνεται στη Λιβύη και διαπιστώνοντας ε, ποια είναι η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα πράγματα μπορούν να σοκάρουν πολλούς από εμά. Είναι φοβερά πράγματα όλα αυτά διότι δεν προχωράν ποτέ. Και όταν εσείς αναφέρατε τις 8 συμβάσεις. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έφυγε ακόμα από τη ΔΟΕ όταν έχει υπογράψει τη συνθήκη της Λισαβόνας. Στην πρώτη μου έκθεση εδώ σε αυτήν την Επιτροπή, είτε πρόκειται για το, MEDA, για το πρόγραμμα ΜΕΝΤΑ είτε για την, ε, την Ισία, αφορούσε στη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτή τη χώρα, είναι το άρθρο 2, που όλοι το ξέρουν ε, από μνήμης που μιλάει για δικαιώματα του ανθρώπου κλπ. Αλλά φαίνεται ότι αποτελούσε αγένεια να χρησιμοποιήσουμε αυτό το άρθρο 2 και να το εφαρμόσουμε, πόσο μάλλον δηλαδή και όταν τα δικαιώματα των ανθρώπων, ε, τα δικαιώματα συγγνώμη των γυναικών δεν ε, ήταν απόλυτα σεβαστά κλπ. Πρόκειται για κάτι το ιδιαίτερα μακρόπνο, βέβαια δεν πρέπει εμείς να σταματήσουμε να, να χαμηλώσουμε την ε, επαγρύπνησή μας, αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Λιβύη είναι φοβερά πράγματα. και οι συνάδελφοι συνεισέφεραν στη συζήτηση πηγαίνοντας προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι τώρα βέβαια 155 είναι αυτές οι 155 τροπολογίες οι οποίες δεν νομίζω ότι αμφισβητούν την αρχική εργασία αλλά απλώς αποδεικνύουν ε, και το ενδιαφέρον ε, της Επιτροπής για τα θέματα αυτά. Εγώ εδώ δεν ε, ρίχνω, βάζω κερασάκι πάνω στην τούρτα. Τώρα, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν θέλει το λόγο. Ναι να απαντήσετε και στην ερώτηση του κυρίου Χάουιτ για το ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λέγομαι Σρέμπερ και είμαι ε, από την ε, υπηρεσία που ασχολείται με διεύρυνση και κοινωνικά θέματα και πολιτική γυτνίασης. Εν γέννη είναι πολλές οι τροπολογίες θα έλεγα και μπορώ να καλωσορίσω κάποιες τροπολογίες διότι διευκρινίζουν ζητήματα και αυτό είναι χρήσιμο κατά τη γνώμη μας η αναφορά ε, στη δήλωση του 2008 για την ε, κοινωνική δικαιοσύνη και τη δίκαιη παγκοσμιοποίηση από τη ΔΟΕ παραδείγματος χάρη, τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, ε, τα περί κοινωνικής εταιρικής ευθύνης του κυρίου Χάουιτ, νομίζω ότι συμπληρώνουν την έκθεση με πολύ ωραίο τρόπο. Για την ΔΟΕ, Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες που τονίζουν το ρόλο της οργάνωσης και των εργασιών που επιτελεί. Πέντε, ζητήματα, αν μου επιτρέπετε, θέλω να σχολιάσω. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη το πρώτο. Ε, γνωρίζετε κύριε Χάουιτ, γιατί έχουμε συνεργαστεί επί μακρόν στο παρελθόν, ότι είμαστε αφοσιωμένοι και θέλουμε να προωθήσουμε την εταιρική κοινωνική ευθύνη ώστε να ε, συμμορφώνονται επιχειρήσεις με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για αυτό το θέμα. Επίση, έτσι ασχολούνται και οι δημοσίε αρχέ με την προστασία των βασικών δικαιωμάτων και είδατε ε, τα περικρατικών προμηθειών και την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ε, επίσης, συμβάλλουμε στη διαδικασία που ανέφερε και ο κύριος Σαχαρίτε για τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ για τις πολυεθνικές και αυτό είναι η συνέχεια της δράσης του επικεφαλής για τα θέματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα επίσης ε, ε, για την εταιρική κοινωνική ευθύνη να σας πω ότι προετοιμάζουμε μια νέα ανακοίνωση για αυτό το θέμα η οποία θα βασιστεί στην εθελούσια μέθοδο που επιλέξαμε το 2006 αλλά ε, δεν θα αποκλεί και άλλου τύπου δράσεις. Ο ορισμός της εταιρική κοινωνική ευθύνης, η υποβολή εκθέσεων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λογοδοσία και ρεσιμότητα για τις επιχειρήσεις μερικά από τα στοιχεία που θα συμπεριλαμβάνει η ανακοίνωση. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πότε θα δημοσιευθεί, αλλά ε, είναι η κοινή πρωτοβουλία των Επιτρόπων στην οποία αναφερθήκατε δεν μπορώ να αναλάβω συγκεκριμένη δέσμευση για την ημερομηνία, νομίζω μετά το καλοκαίρι, αλλά ε, συνεχίζει τη συνεργασία των Επιτρόπων. Για το θέμα των διεθνών προτύπων, ε, προφανώς ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Τα εργασιακά πρότυπα του, της ΔΟΕ είναι ήδη ενσωματωμένα στις εμπορικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα σχετιστούν με το κεφάλαιο περιβιώσιμης ανάπτυξης που περιέχει κάθε νέα συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών. Ε, αυτό το επιδιώκουμε σε όλες τις σχέσεις που έχουμε με τρίτες χώρες μέσω αυτών των συμφωνίων συμφωνιών και θέλουμε οι εταιροί μας να διατηρήσουν τις προσπάθειές τους ούτως ώστε να εφαρμόσουν τις ε, συμβάσεις ε, που, έχει εκδώσει, ε, που έχουν προσπογράψει γνώμη με την ΕΔΟΕ. Δεν μπορούμε φυσικά να υποχρεώσουμε τους εταίρους μας να το κάνουν αυτό, αλλά μπορούμε να ασκήσουμε πίεση επίσης. Απαιτούμε μια αυξημένη δέσμευση και αποφόσιωση από πλευρά των χωρών εταίρων. Δεν έχετε τη βασική αρμοδιότητα βέβαια για τη διαπράγματευση των εμπορικών συμφωνιών, αλλά πάντως θα γνωρίζετε ότι χρησιμοποιούμε αυτό το μέσο πίεσης ε, στις σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες, ε, κυρίως όταν διαπραγματευόμαστε νέες συμφωνίες. Μους χρειαζόμαστε όμως και κάποιο μέτρο σύγκρισης ε, πριν προχωρήσουμε. Η γραμμή μας μέχρι τούδε είναι ότι εάν γίνει αυτό θα έχουμε μικρότερη μόχλευση, μικρότερη πίεση μπορούμε να ασκήσουμε ε, στα κράτη-μέλη. Και μην ξεχνάτε ε, ότι μπορεί θεωρητικά να είναι καλύτερο να έχουμε ένα μέτρο σύγκριση πριν ξεκινήσουμε τι διαπραγματεύσει. Στην πράξη είναι διαφορετικά τα πράγματα. Κατόπιν αυτή η πρόταση για ένα νέο κανονισμό για τις γενικευμένες προτιμήσεις ε, που θα ε, κατατεθεί το 2011, νομίζω έχουμε χρόνο για να επανέλθουμε. Για την ε, Μεσόγειο προφανώς παρακολουθούμε στενά το ζήτημα και στο παρελθόν έχουμε ξεκινήσει περιφερειακό διάλογο με τις μεσογειακές χώρες και έχουμε συγκροτήσει και ένα φόρουμ κοινωνικού διαλόγου με βασικούς εταίρους μας όπου συζητούμε πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα, ζητήματα που σχετίζονται με τις δεξιότητες, τα προσόντα, την αναγνώριση αυτών. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε τώρα είναι ε, να ε, βοηθήσουμε τα νέα συνδικάτα ε, και να συνεργαστούμε με κυβερνητικέ οργανώσεις. Και... Πρέπει να δούμε στο Κοινοβούλιο ότι πραγματικά μπορούμε να έχουμε μια λογική καλή δέσμευση already, για να δούμε τι έχουμε κάνει, πώς έχουμε γνωρίσει τα διάφορα θέματα. Αυτό ε, το θέμα της ανεργίας των γυναικών, παραδείγματος χάνει όλα αυτά τα σχετικά πρόβλημα. Θα είδατε σίγουρα την ε, ανακοίνωση της Κομισιόν ε, που υιοθέτησε η πατός εκπρόσωπος όσον αφορά το θέμα της ε, συμφωνίας ε, με την Μεσόγειο. Πολλά θέματα που θα πρέπει να υποστηρίξουμε όσον αφορά τις δημοκρατικές μεταβάσεις. Προσπαθούμε στο δικό μας τομέα να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και τελειώντα, κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε στην ομάδα των 20 στο G20. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Κομισιόν υποστηρίζει τη Γαλλική Προεδρία για το θέμα αυτό και μπορούμε πολλά να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής πώ θέλει να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Já jsem nechtěl kolegyně a kolegy postrašit řadu pozměňovacích návrhů. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ δεν θέλω να τρομοκρατήσω τους συναδέλφους. Εγώ προσπάθησα απλώς να εκφράσω τη θέση μου. Και το λέω αυτό απευθυνόμενος ε, στην ε, Κομισιόν. Μα εμένα μου φαίνεται ότι περάσατε τα τελευταία πέντε χρόνια σε έναν άλλο πλανήτη. Ο Επίτροπος Πίτλα τότε είχε προτείνει μια οδηγία που δεν πέρασε από το Κοινοβούλιο για το ωράριο εργασία. Αλλά τέλος πάντων κάποια επικοινωνία θα πρέπει να είχατε και με, με τις αφρικανικές χώρες δεδομένου και της κατάστασης σήμερα. Και χαίρομαι που δεν ακούστηκαν πολλές κριτικές. <laughs> Αλλά στον συνάδελφο Χάουιτ λέω το εξής. Σύμφωνο σε μεγάλο βαθμό με τις τροπολογίες του και σε μεγάλο βαθμό και με τις τροπολογίες της Προέδρου. Δηλαδή εγώ δεν διαμαρτύρομαι για να διαμαρτύρομαι. Κοιτάξτε αυτό είναι και το ενδιαφέρον μιας έκθεσης ε, πρωτοβουλίας αυτόν τον τομέα. Ε, θέλει να περάσει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων μερικά ισχυρά μηνύματα ας πούμε για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων θα πρέπει να προχωρήσουμε αν δούμε δηλαδή και αυτή την τελευταία ψηφοφορία που έγινε και τα λοιπά μπορούμε να έχουμε μόνο πλεονεκτήματα η έκθεσή σας κύριε Φάλμπρα τον Απρίλιο θα συζητηθεί Πρέπει όμως να βρεθούμε για να συζητήσουμε τις συμβιβαστικέ τροπολογίες, διότι θα τις έχετε ήδη προτείνει. Πάμε τώρα στο 34. Πόσο μάλλον επίκαιρο το θέμα. Όχι βέβαια στην Ήπειρό μας, αλλά εξίσου δύσκολο όμως. Η κυρία Τζιν Λάμπερτ για τη γνωμοδότησή σας για την Ήτρε για τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως είπατε, το θέμα αυτό είναι άμεσο ενδιαφέροντος. Θα προτιμούσαμε βέβαια να έχουμε τη ζήτηση κάτω από διαφορετικές προϋποθέσεις. Από την άλλη μεριά είναι σαφές ότι έχουμε πολλές παρουσιάσεις στα ΜΜΕ που παρουσιάζουν τα προβλήματα της χειρότερης δυνατής περίπτωσης. Και όλες αυτές οι εκθέσεις μεταξύ άλλων αναφέρονται στις επιπτώσεις στους εργαζομένους στην Ιαπωνία, του Φουξίμα. Και κοιτάμε πώς το αντιμετωπίζουν με την χρήση των ε, εργαζομένων ε, κυκλικά για να μην εκτίθενται σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας. Η έκθεση που εξετάζουμε στην Επιτροπή μας εντάσσεται στη συζήτηση που γίνεται στην Επιτροπή Ήτρε αυτή τη στιγμή. Η πρώτε οδηγίε είναι μέσα στα πλαίσια της συνθήκη Ευρατών. Και γι' αυτό ε, ζητάτε να γνωμοδοτήσουμε. Η υποστηρικτική αιτιολόγηση της Επιτροπής αναφέρει τη βασική αργή της διαχείρισης διαδημιουργών αποβλήτων περιλαμβάνει τον περιορισμό και την απομόνωση από του ανθρώπου και την βιοσφαίρα για όσο διάστημα αυτά συνιστούν ραδιολογικό κίνδυνο. Επιπλέον, α, αναφέρεται ότι πρέπει η σημερινή κοινωνία να ε, διαχειριστεί σωστά τα υπάρχοντα απόβλητα. Αυτό είναι το σημείο της ε, αδική μας πρότασης. Εξετάσαμε δηλαδή να διευρύνουμε τις πτυχές για να καλύπτουμε την υγεία και την ασφάλεια, να εξετάσουμε δηλαδή, τους εργαζομένους σε όλη την αλυσίδα της ε, χρήσης, ε, της αντιμετώπισης αν θέλετε των αποβλήτων αυτών, όχι μόνο τους ειδικού, αλλά οποιοδήποτε ακόμα και οι ε, δυνάμεις ασφαλείας, εκείνοι που κατά σύπτωση εργάζονται με αυτό, εκείνους που έχουν αναλάβει υπεργολαβίες κλπ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για χώρες όπως ε, τη δική μου. Εξάζουμε με τα θέματα της προστασίας, της εκπαίδευσης και να εξετάζουμε τι καλύπτεται, τι σημαίνει δηλαδή ε, κατά βάση ε, απόλυτο και αναλωμένο καύσιμο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες, πολλές από τις οποίες μπορώ να υποστηρίξω. Σε ορισμένες ίσως θα ήταν καλό να συζητήσω με τον, υποβα... τον υποβάλλοντα ε, κατά πόσον η διατύπωση είναι ιδανική, αλλά γενικά πραγματικά τις περισσότερες μπορώ να τις υποστηρίξω. Και υπάρχουν και ορισμένες χρήσιμες νέες ιδέες που έχουν υποβληθεί μέσα στα πλαίσια αυτών των τροπολογιών. Ιδίω όσον αφορά την ανάγκη να κρατούνται κατάστοιχα όπω η 19 του κ. Χάντα για το 6-2 δέλτα νέο. Και το θέμα ότι πώς ε, παρακολουθούμε τους εργαζόμενους σε ο οποιαδήποτε ε, δραστηριότητα ε, δημιουργεί απόβλητα ραδιενεργά, όπως παραδείγματος χάρη είναι στο νοσοκομείο που είναι χαμηλής με ραδιενέργειες, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να τους παρακολουθήσουμε. Έχω κάποιες ε, ερωτήσεις. Η μία αφορά τη νομική βάση. Η αρχική μου πρόταση είχε προτείνει να αλλάξει η νομική βάση από το, τη συνθήκη Ευρατών στο άρθρο 153 της συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την δημιουργία των προτύπων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Οι τροπολογίες 42, 43, 44 σχετίζονται με την Ευρατόμ και επίσης και 40 και 46 που αναφέρεται σε μια κοινή νομική βάση. Είναι κάπως προβληματικές δηλαδή, γιατί βλέπουμε δύο διαφορετικούς μηχανισμούς λήψης απόφαση. Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες, ιδίως κυρία Πόμ, για το θέμα των εξαιρέσεων μέσα στα πλαίσια της οδηγίας. όσον αφορά συγκεκριμένες ε, μορφές διενεργών δηλαδή αποβλήτων όπως εκείνα παραδείγματος από την εξόριξη του ουρανίου. Γι' αυτό οι τροπολογίες μου 13 και 14 προβλέπουν να εξελθούν αυτές οι εξαιρέσεις. Καταλαβαίνω βέβαια ότι μία από τις οδηγίες που αναφέρονται η 2021 σχετίζεται με την εξόρυξη δεν επισέρχεται στις ε, λεπτομέρειες και στα πρότυπα εργασίας για τους εργαζόμενους. Άλλο θέμα αφορά το χρονοδιάγραμμα. Μέχρι πότε δηλαδή θα πρέπει να ασχοληθούμε με κάποια συγκεκριμένα θέματα και κάποιες τροπολογίες, η 17 Φερρυπίν, λένε ότι εντάξει, ας κοιτάξουμε έναν ορίζοντα 150 ετών. γιατί ορισμένα από τα υλικά αυτά έχουν ε, που, αυτή τη διάρκεια ζωής, άλλα όμως έχουν μεγαλύτερο διάστημα ακτινοβολίας και μετά έχουμε τις ε, τροπολογίες 34-35 που παρατείνουν αυτή την πρόταση και προβλέπουν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Ελπίζω να ακούσω κάποια σχόλια για αυτό και υπάρχουν διάφορα σημεία του κειμένου όπου θα πρέπει να αποφασίσουμε ποια είναι η καλύτερη διατύπωση. Θεωρώ παραδείγματο χάρη ότι η τροπολογία 80 της κυρίας Στάνλο και που αναφέρεται στην νομική βάση είναι καλύτερη από τη δική μου και την τριαδανία του κ. Χάνλο. Όσον αφορά στι συμβαστικέ ε, τροπολογίε ενδεχόμενα, νομίζω ότι πολλέ από τι τροπολογίε είναι πολύ ξεκάθαρε. Αλλά το άρθρο 9 θα μπορεί νομίζω να ξαναεξαρθεί και να βρούμε ένα συμβαστικό κείμενο. Γι' αυτό καθώς επίσης και για το 6.3 που αφορά το εθνικό πλαίσιο. Είπαμε το 9 και το 6.3 είναι δύο άρθρα για τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε σε συμβαστικές τροπολογίες, είμαι σίγουρη. Και από τις τροπολογίες που έχουν βιβλίο πολλές μπορούν να δεχτώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε κύριο Στάινφρικ, ευχαριστώ την Τζιν Είχαμε ξανασυζητήσει την έκθεση αυτή. Είναι πάρα πολύ καλή νομίζω. Οι τροπολογίε ε, δείχνουν ότι κινούνται προ την ίδια κατεύθυνση. Ε, δυναμώνουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Και για να απαντήσω ε, κάποιε ερωτήσει που υπευλήθησαν σχετικά με τι τροπολογίε μου, έχω να πω ότι για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό η οδηγία να τοποθετηθεί σε ευρία νομική βάση για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε έτσι την ασφάλεια νομικής βάσης, ιδίως όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων. Νομίζω ότι μπορούμε ξανά να συζητήσουμε στις λεπτομέρειες τις διάφορες νομικές βάσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει, όχι μας μόνο στους ελιστές αλλά όλους, είναι ε, το θέμα της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας όσον αφορά και τις στρατιωτικέ χρήσεις. Αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να εξεράσουμε κάποιους βιομηχανικούς τομείς για τους οποίους μετά δεν θα υπήρχε καμία βάση για την προστασία της εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος και της υγείας χρειαζόμαστε επαρκές αρμοδιότητες ε, της διακανοστικής αρχής. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι η οδηγία να επιτρέπει στα κράτη-μέλη να υπάρχουν υψηλότερα πρότυπα. Αυτό είναι κάτι με το οποίο είχαμε κακές εμπειρίες σε άλλους τομείς. Αλλά ακριβώς συζήτησα το θέμα στη Γερμανία με διάφορες οργανώσεις και επιχειρήσεις και ξέρω ότι εν μέρει υπάρχουν πολύ υψηλότερα πρότυπα και υπήρχε ο φόβος ότι εμείς θα μειώσουμε τα πρότυπα αυτά, όπως το έχουμε κάνει και σε άλλους τομείς. Και έχω και μία ερώτηση προς τον κύριο Σόγκαρ, ο οποίος σε μία τροπολογία προβλέπει υποστήριξη εκείνων που έχουν στα χέρια τους ε, κάποια άδεια ε, τι εννοείται, εννοείται οικονομική υποστήριξη, αυτό θα με προβλημάτισε. Ε, τι εννοείται, τέλο πάντων μπορούμε μετά να το συζητήσουμε και μεταξύ μα. Είμαι σίγουρο ότι θα έχουμε πολύ καλές ε, συζητήσεις και ακριβώς αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε ένα καλό αποτέλεσμα και ομόφωνο στην αποτελεσματική γνωμοδότηση μας προς την Επιτροπή Ήτρε γιατί θα πρέπει να προσπαθήσουμε μην ξεχνάμε ποια είναι η έκθεση των ατόμων που εργάζονται με τι ουσίε αυτέ, ιδίω βλέποντα την επικαιρότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χρειάζεται πραγματικά ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, γιατί πρέπει να ξεχνάμε τον ανθρώπινο παράγοντα που μπορεί να ασφαλεί και δεν πρέπει να ξεχνάμε τις μελλοντικέ γενιές. Και γι' αυτό υπάρχουν τόσες πολλές τροπολογίες. Ε, σε μερικέ διαφέρουμε. Δηλαδή, εμείς δεν θέλαμε να αναφέρουμε συγκεκριμένο αριθμό ετών πόσα χρόνια θέλουμε να φροντίσουμε για την ασφάλεια. Δηλαδή να πούμε 250 χρόνια και τελείωσε. Όχι. Θα πρέπει να δούμε ε, την διάρκεια της ε, ε, ραδιενεργούς ακτινοβολίας των ε, ε ουσιών αυτών. Υπάρχουν πολλές ε, τροπολογίες που επικαλύπτουν. Θα τις τη με τους συναδέλφους και δεν νομίζω θα υπάρχουν προβλήματα. Αυτά ήθελα να προσθέσω και θα ήθελα να ευχαριστήσω για την έκθεση την εισηγήτρια και θεωρώ ότι είναι πολύ καλό να μην ξεχνάμε ότι αφενός χρειαζόμαστε την πυρηνική ενέργεια, από την άλλη μεριό μας χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί για να μπορέσουμε να ε, χειριστούμε σωστά τα ραδιενεργά απολοπόβλητα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και ε, ένα κυριαρχικό δικαίωμα ενό κράτου μέλου να χρησιμοποιεί την ε, ραδιενέργεια και για παραγωγή ενέργειας και για ιατρικούς λόγους, αλλά κάθε κράτος θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες προστασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να πω ότι πραγματικά εντυπωσιάστηκα στο πόσες τροπολογίες έχουν κατατεθεί. Ε, πρέπει να... Πρέπει σίγουρα να γνωμοδοτεί η Επιτροπή ε, απασχόλησης αλλά από την άλλη μεριά όταν βλέπουμε το πώς μεταχειρίζονται τις ε, γνωμοδοτήσεις στις αρμόδιες επί της ουσίας επιτροπές ε, νομίζω και εμείς δηλαδή θα πρέπει κάπου να μετριάσουμε τη δράση μας και να ασχολούμαστε, να, να περιορίζουμε το πεδίο μόνο στις ε, αρμοδιότητες της Επιτροπής μας, απασχόληση και κοινωνικά θέματα. Δείτε το πακέτο για την ευκυβερνησία που κατέληξε, που θεωρήθηκαν απαράδεκτες αρκετές τροπολογίες γιατί ήταν εκτός θέματος. Πρέπει λοιπόν να είμαστε αποτελεσματικοί. Η κυρία Λαμπέρτ θέλει να συνεχίσει. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους αδέλφους για τα σχόλιά τους. Όπω είπε και ο κ. Σόκορ, πραγματικά υπάρχουν ορισμένε τροπολογίε που είναι παρόμοιε, που καλύπτονται και μπορούμε να δούμε ποιε θα είναι εκείνε τελικά που θα υπάρχουν στον κατάλογο ψηφοφορία. Το θέμα της ε, του μήκους μιας γνωμοδότησης. Ε, δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι ε, είναι περιοριστικό. Προσπαθήσαμε να το ακολουθήσουμε γιατί είναι και θέμα του τι μας απασχολεί. Um, Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φροντίσουμε ε, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε εδώ ένα νομικό κείμενο και Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα κρατήσει από αυτά που θα πούμε η επί αρμόδια επιτροπή. Πάντως προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε κάποια σημεία. Υπήρξαν επικρίσεις σήμερα γιατί επέκρινε κάποιος στην εργασία άλλων θεσμικών οργάνων. Δεν θα πω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ τους συναδέλφους πάντως για τα σχόλιά τους. Ε, Οι άλλες επιτροπές ε, συμφωνούν να κρατούν τις νομοδοτήσεις ε, και πολλές φορές κινητοποιούν και τους προέδρους τους για να επηρεάσουν την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όταν εμείς εγκρίνουμε την εισήγηση, ο εισηγητής να μπορεί να το προχωράει μέχρι το τέλος. Πάμε τώρα στις διαδικασίες αφαιρεγγιότητας στο πλαίσιο της νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιχειρήσεις. Η κυρία Ζουλή Γκίρλινγκ Α, ξέχασα το χρονοδιάγραμμα για την έκθεση της κυρίας Λαμπέρ. Για την έκθεση της κυρίας Λαμπέρ, η έκθεση των συμβιβαστικών τροπολογιών θα γίνει στις 13 Απριλίου και θα ψηφίσουμε στις 14. Η κυρία Γκίρλινγκ για τις διαδικασίες αφαιρεγγιότητας και λοιπά για την νομική επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπό το φως ε, των παρατηρήσεων που μόλις κάνατε για τις ε, γνωμοδοτήσεις ε, και τις τροπολογίες, νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα και ελπίζω να μην έχουμε υπερβολικά πολλές τροπολογίες η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θέλησε να διερευνήσει περαιτέρω την εναρμόνιση ε, στο τομέα ε, της αφαιρεγγιότητας, ε, κυρίως στη διοικητική δικαστική διάσταση του ζητήματος και εξέδωσε το σχέδιο έκθεσης Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Δεν ασχολούνται βέβαια με την διάσταση της απασχόλησης, θέμα που θα εξετάσω εγώ στη γνωμοδότησή μου. Το συμπέρασμα μου είναι ότι η οδηγία του 2008 που επιθυμούν να τροποποιήσουν τώρα από πλευρά κοινωνικών υποθέσεων και απασχόληση έχει λειτουργήσει αισίω ε, και είναι δύσκολο να πιστούμε για την ε, χρησιμότητα της ε, τροποποίησης. Προσπάθησα πραγματικά ε, μέσα στον κανονισμό του 2008 για την ε, αφαιρεγγιότητα να εντοπίσω σημεία που θα έπρεπε να αλλάξουν, ε, αλλά δεν ε, εντόπισα πολλά τέτοια σημεία. Το γενικό μου συμπέρασμα ε, θα είναι να μην κάνουμε αλλαγές όταν λειτουργεί αισίως το σύστημα από πλευράς απασχόλησης. Ε, έλαβα υπόψη την ε, άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Κοινωνικών Εταίρων και υπάρχει ευρεία συνένεση σχετικά με το ότι λειτουργεί ικανοποιητικά ο κανονισμός του 2008. Προσπάθησα να εξετάσω και το θέμα τη επικουρικότητας και της ευελιξίας των κρατών μελών Φυσικά είναι σημαντικά αυτά τα ζητήματα, αλλά θέλω όλα να είναι απλά. Δεν θέλω να υπερβάλλω υπέρμετρα ένα νομοθέτημα που λειτουργεί ούτως ή άλλως ε, ικανοποιητικά. Θα ήθελα να ακούσω απόψεις για ένα θέμα που ακόμη, ε, για το οποίο μάλλον δεν έχω καταλήξει. Ε, δηλαδή, θα ήταν δυνατόν να ε, προκύψει μια νομοθετική πρόταση με θετικό αντίκτυπο σχετικά με ε, την, ε, αυτό που ονομάζουμε τουρισμό αφαιρεγγιότητας, δηλαδή διαλέγουν οι εργαζόμενοι ποια είναι κατάλληλη χώρα για αυτούς, ούτως ώστε να δηλώσουν αφαιρέγγι και να κηρύξουν πτώχευση. Το θέμα της απασχόλησης έχει αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ιεραρχική, αν θέλετε, κατάταξη των επιστοτών και αυτή η ιεραρχία φυσικά ε, καθορίζει τον τρόπο αποζημίωση σε περίπτωση πτώχευσης. Ε, αυτό είναι το θέμα που μα ενδιαφέρει περισσότερο από πλευράς απασχόλησης και θέλω να ακούσω και την ε, άποψη των συναδέλφων. Ευχαριστούμε, η κυρία Μοχά. Εγώ θα θα, εκπρα... θα, θα εκπροσωπήσω τον Φιλίπ ο οποίος είναι και ο σκιώδης εισηγητής για το ΕΛΚ και ο οποίος ε, δεν μπόρεσε να μείνει μέχρι τώρα. Ζητά λοιπόν συγγνώμη. Ο κύριος ε, Μπουλά ε, ευχαριστεί την κυρία Γκέρλινγκ για το θέμα της αφαιρεγγιότητας Αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει ε, ε, να επανεξετάζονται μάλλον στην αποτίμηση της εφαρμοστικής τους ε, φάσης και αυτό μέσα σε ένα πλαίσιο σε ένα πλαίσιο παγκόσμιας κρίσης. Εμείς ως ΕΛΚ θα το δούμε επικοδομητικά το θέμα και όπου θα συνδυάσουμε τις κοινωνικές ευθύνες Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επικουρικότητα των κρατών μελών. Θα δούμε το θέμα των πιστωτών, των επιχειρήσεων, των εγγύσεων και την συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Επίσης, επίπεδο επιχειρήσεων ε, θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να παλέψουμε κατά της ε, ε, διακίνησης των, των ταμείων και χρημάτων κινητών και κινήτων των επιχειρήσεων μέσα στην Ένωση. Εμείς θέλουμε να πετύχουμε μια μεγάλη συνένεση γύρω από τα σημεία 3, 4, 8 και 9 όπου η προσέγγιση μας είναι πιο ε, διαφοροποιείται και θα προτείνουμε τροπολογίες. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ την εισηγήτρια για τις προτάσεις και θα σταθώ σε ένα από τα σημεία τα οποία αναφέρθηκε είναι το θέμα της πτώχευσης στον τομέα του τουρισμού. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εμείς με το θέμα του επιχειρησιακού δικαίου διότι όλα αυτά πολλές φορές καλύπτονται και με τη μετατόπιση των επιχειρήσεων. Όπως είπε και η προλαλήσασα, όλα πάνε προς την καλή κατεύθυνση Και φυσικά εμείς θα καταθέσουμε τροπολογίες με την καλύτερη συνεργασία με την εισηγήτρια. Κανένας άλλος θέλει το λόγο, όχι. Εγώ να προσθέσω μία παρατήρηση, δεν ξέρω ποιες θα είναι οι τροπολογίες που θα καταθέσουν οι συνάδελφοι, αλλά αν εμείς πρέπει να ε, παλέψουμε κατά της αφαιρεγγιότητας, δεν, στον τομέα του τουρισμού δεν μπορούμε εμείς να αγνοήσουμε και το θέμα των εγγύσεων. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτή τη θεματική όταν θα έχουμε τις τροπολογίες μέχρι τις 22 Μαρτίου. 14 Απριλίου θα ψηφίσουμε και η Νομική Επιτροπή θα ψηφίσει στις 23 Ιουνίου. Τελευταίο σημείο τώρα στην ημερήσια διάταξη και ευχαριστώ τους συναδέλφους που έμειναν μέχρι το τέλος. Πρόκειται για ένα θέμα στο οποίο πρέπει προφορική ερώτηση μάλλον για, με ψήφισμα σχετικά με τη σύμβαση της ΔΟΕ για τους οικιακούς βοηθούς. Λοιπόν, έχει συνταχθεί προφορική ερώτηση, πρέπει να ανοιχτή για να μαζέψει υπογραφές και θα συζητηθεί την Τρίτη και την Τετάρτη το θέμα και στη Γενέβη με προσώπους της ΔΟΕ και τον Γενικό της Διευθυντή. Θέλετε εσείς κάποια αλλαγή για την προφορική ερώτηση και για το σχέδιο ψηφίσματος. Υπάρχουν αντιδράσεις ή θέλετε να περιμένουμε τη Γενέβη για να εμπλουτίσουμε και την ε, σκέψη μας. Εγώ νομίζω ότι η αρχή που ενέκριναν οι συντονιστές ήταν ε, ομοφωνία. Τώρα να δούμε βέβαια πώς θα τα εμπλουτίσουμε όλα αυτά μετά από την, επιστροφή μας στη Γενέβη. Ε, κυρία Μωρά. Κυρία Πρόεδρε, εμείς συμφωνούμε με αυτό το κείμενο έτσι όπως το είχαμε ήδη προσυμφωνήσει και, στην, και στους συντονιστές και θα περιμένουμε τη Γενέβη ούτως ώστε μετά να μπορέσουμε να εντάξουμε και τον καρπό των συζητήσεων. Θα ήταν πρόωρο να κάνουμε οτιδήποτε σήμερα. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, λέει ο κύριος Θέρκας χωρίς μικρόφωνο, μικρόφωνο κύριε Θέρκας. Να πάρω άλλο, αυτό δεν δουλεύει. Εγώ πάντα παίρνω το μικρόφωνο από αριστερά, ενώ πρέπει να το παίρνω από δεξιά τελικά. Έλεγα λοιπόν, Πρόεδρε, ότι συμφωνώ απόλυτα με τη συνάδελφο του ΕΛΚΑ. Πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο το αποφασίσαμε στην, ε, στους συντονιστές, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και την ε, τύχη να γνωρίζουμε πολύ καλά το τι σκοπεύουν να συζητήσουν στη Γενέβη. Η συζήτηση θα είναι πολύ πλούσια όταν γυρίσουμε από τη Γενέβη. Και μπορούμε λοιπόν τότε να συζητήσουμε το κείμενο σε μια επόμενη συνεδρίαση. Εκπρόσωπος της Κομισιόν θέλει να πει κάτι. Όχι για να σχολιάσει την ποιότητα της πρωτοβουλίας, αλλά απλώς για να συνεισφέρει στο θέμα της υπογραφής αυτής της σύμβασης. Ε, Βεβαίω, μπορώ να σας δώσω κάποιες γενικές ε, πληροφορίες, αν το επιθυμείτε. Ωραία. Αφού συμφωνείτε, θα επαναλάβω τη σημασία που ε, προσδίδουμε στο θεματολόγιο για την αξιοπρεπή εργασία. Ε, ανέκαθεν παρακολουθούσαμε στενά και διευκολύναμε το συντονισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη για τις συμβάσεις ε, που έχουν εγκριθεί, τις συμβάσεις της ΔΟΕ. Δηλαδή, επίσης, θα συζητήσουμε και στο μέλλον την ε, προσέγγιση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Ε, το 2010 έγινε διεθνή διάσκεψη για τα εργασιακά ζητήματα, ειδικοί, αξιωματούχοι του ΔΟΕ συμμετείχαν στη διάσκεψη και όπως και οι συμβάσεις που είχαμε διαπραγματευτεί τα περασμένα χρόνια, ε, οδηγηθήκαμε σε εξέταση των διαθέσιμων εργαλείων ε, και τον παραλληλισμό με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, για ποιο λόγο, διότι εγκαίρως θέλουμε να εντοπίσουμε τα σημεία όπου υπάρχει τυχόν θέμα συμβατότητας με το κεκτημένο της Ένωσης και μετά εξετάζουμε το περιεχόμενο των νομικών πράξεων του κεκτημένου που εντοπίζουμε το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η νέα σύμβαση της ε, ΔΟΕ θα καλύπτει και θέματα αρμοδιότητας ε, της Ένωσης. Ε, προφανώς τα κράτη-μέλη πρέπει να τηρούν το κεκτημένο, αλλά σε πολλούς τομείς, θα το ξέρετε, προβλέπονται ελάχιστα πρότυπα μέσα στο κεκτημένο και τα κράτη-μέλη προφανώς έχουν τη διακριτική ευχέρεια να δεχτούν και να επικυρώσουν διεθνή μέσα, παρέχοντας έτσι υψηλή προστασία. Τα πρότυπα βέβαια της ΔΟΕ προβλέπουν αυτά τα ελάχιστα πρότυπα, άρα θα πρέπει να διατηρηθεί το κεκτημένο, να προστατευτεί από τα κράτη-μέλη και είναι σημαντικό να το τονίσουμε. Για τον επόμενο και αποφασιστικό γύρο συζητήσεων στη Διεθνή Διάσκεψη Εργασία θα συνεχίσουμε να έχουμε ενεργό ρόλο και να διευκολύνουμε τα κράτη-μέλη, τόσο να γίνεται εγκαίρωση ε, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ειδικών, μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων και θα συνεργαστούμε φυσικά και με τον εισηγητή τη οικονομική και Κοινωνικής ε, σχετικά με την τον επαγγελματικό χαρακτήρα της εργασίας των ε, οικιακών βοηθών. Αυτά, με αυτά ασχολούμαστε. Ας περάσω και στην ουσία. Ο πλευρά απασχόληση, προφανώ υποστηρίζουμε αυτό το ε, στόχο σχετικά με το προφίλ των οικιακών βοηθών και θα θέλαμε, δεδομένου των δημογραφικών εξελίξεων και τη αυξημένη συμμετοχή στην αγορά εργασία από πλευρά των γυναικών, να κάνουμε τι απαιτούμενε προσαρμογέ, αλλά φυσικά ε, θα πρέπει να εφαρμόσει τα πρότυπα της ΔΟΕ ε, για τους ε, οικιακούς βοηθούς. Μιλήσατε για την επισφαλή θέση στην οποία βρίσκονται αυτοί οι εργαζόμενοι. Θα πρέπει, πιστεύουμε, να θεωρούνται όλοι ως κατέχοντες μια επισφαλή θέση εργασίας και μετά να περάσουμε στον προσδιορισμό του προφίλ αυτών των βοηθών και σε διάφορα κράτη έχουμε σχετικές εμπειρίες σε αυτή την ε, απόπειρα να ε, αμβλύνουμε κάπως τον επισφαλή χαρακτήρα αυτής της απασχόλησης. Να σας δώσω και συγκεκριμένα παραδείγματα. Ε, υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα, το παραδείγμα χάρη, που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα το υλοποιούμε, που ενθαρρύνει τη σύγκληση ή μάλλον το πέρασμα από την επισφαλή θέση απασχόληση, μια που γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γίνεται και μια μελέτη Μάλλον θα γίνει μια μελέτη πέρα από το πιλωτικό πρόγραμμα για να εξεταστεί αυτό το φαινόμενο των επισφαλών θέσεων εργασία όλη την επικράτεια της Ένωσης για να επιτύχουμε αυτό το πέρασμα από τις επισφαλείς θέσεις, ε, κατογερωμένες με συμβάσεις ε, και προστατευμένες θέσεις εργασίας σε συνδυασμό με τα εθνικά μέτρα που έχουν φυσικά τον ίδιο στόχο, περνώντας από την ε, αναγνώριση των αδυναμιών και των ατελειών σε σχέση με τα κοινωνικά δικαιώματα. Πρόσφατα επίσης ασχοληθήκαμε με την αξιοπρεπή εργασία κάνοντας μια μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων παραβιάζαν των δικαιωμάτων ε, και η μελέτη έγινε στην Ιταλία, δεν ξέρω αν θέλετε λεπτομέρειες, οι συνάδελφοι μπορούν να να σας ενημερώσουν. Αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο. Εάν έχετε τώρα ειδικότερε ερωτήσεις για τη διαδικασία ή για το περιεχόμενο, έχουμε και την ε, νομική δήμον εδώ δίπλα μου, αν θέλει να σας απαντήσει. Τέλεια. Τέλεια. Θα επανέλθουμε στο θέμα αφού θα έχουμε περάσει από τη Γενέβη πρώτα. Τη Δευτέρα και την Τρίτη λέει θα πάμε στη Γενέβη. 24 Μαρτίου προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών στο ψήφισμα στις 5 το απόγευμα. Μόνο αγγλικά. Και έτσι λοιπόν θα Έχετε, θα ψυχαγωγηθείτε στο ταξίδι του γυρισμού γράφοντας τροπολογίες. 13 Απριλίου λοιπόν θα τη συζητήσουμε, 14 Απριλίου θα ψηφίσουμε. Τελειώσαμε. 13-14 Απριλίου. Καλό βράδυ το επόμενο ραντεβού.